Bene, colleghi, se siete d'accordo, iniziamo. Ο πρόεδρο, να αρχίσουμε συνάδελφοι, αν δεν έχετε αντίρρηση. Buongiorno a tutti, do il benvenuto a... Καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε, πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, η Ίγκε Γκρέσλε. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Από πλευρά τη Επιτροπή Γεωργία και Άντρεξη τη Υπαίθρου, ε, την οποία έχω τιμή να εκπροσωπώ, Καλώς ορίσαν όλοι οι σημερινοί και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είναι πολύτιμη συμβολή τους σε αυτήν την κοινή ακρόαση. Έτσι θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε όσον αφορά τη γνώση του leader και θα δούμε πώς ε, μέσα στον χρόνο λειτουργήσε και θα δούμε ποια είναι η προσθέμενη αξία του. Πέραν των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των Κυβερνήσεων, Έχουμε εδώ κάποιους ε, εμπειρογνώμονες, κάποιους ε, ειδικού που ε, ξέρουν πώς λειτουργήσε στην πράξη το leader. Οπότε, θα πρέπει να δούμε τι έγινε στο παρελθόν, αλλά θα πρέπει με αυτή την ευκαιρία να έχουμε κάποια μικρή γνώση για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το leader στο μέλλον. Και όσον αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο σε τα πλαίσια του πι θα δούμε <clears throat> τι θα γίνει. Σε πέντε τμήματα θα διαρθρωθεί η ακρόασή μας. Πρώτα-πρώτα έχουμε τους τρεις ε, εμπειρογνώμονες θα μας μιλήσουν από πλευρά της οργάνων και ε, κυβερνήσεων. Δεύτερο πάνελ, και θα έχουμε τέσσερις ε, ειδικού οι οποίοι θα μας αναπτύξουν την άποψη των εμπλεκομένων. Μετά θα έχουμε ερωταπαντήσεις και τέλος τα συμπεράσματα. Η κάθε παρουσίαση από τους ειδικού ε, θα κρατήσει 10 λεπτά maximum. Και σας τονίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να τηρήσετε αυτό το χρονικό όριο, αυτό το χρονικό περιορισμό. Ωραία. Τώρα. Πρώτο τμήμα της ακρόασης θεσμικά όργανα και κυβερνήσεις. Είπαμε ότι θα ακούσουμε τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία των κυβερνήσεων και των θεσμικών οργάνων και να μας πούν τι γίνεται πριν αρχίσουμε την, ε, η πρόταση της Επιτροπής ε, Λέω προϋπολογισμού πρώτα. Ευχαριστώ και καλωσορίζω και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Μία φορά είχαμε ήδη ε, προγραμματίσει, αλλά τελικά μεταθέσει την ημερομηνία τη σημερινής ακρόαση ε, και να πω εισαγωγικά πως ε, το πρόγραμμα ε, Λίντερ είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, καλύπτει μεγάλο κομμάτι των εκτάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή λειτουργεί διαφορετικά από άλλα προγράμματα γιατί ακριβώ ακολουθεί μια προσέγγιση bottom-up, από τα κάτω δηλαδή προ τα πάνω. Αλλά αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχει και τι δικέ του αδυναμίε. Σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν πολλέ ε, κοινότητε σε τοπικές δράσεις οι οποίε συνδιοργανώνουν το Λίντερ και όχι διοικητικέ αρχέ, η Υπουργεία ή αρμόδιοι οργανισμοί περιφερειακή πολιτική. Άρα λοιπόν εντό εισαγωγικών μιλάμε για εντελώς κανονικούς ανθρώπους οι οποίοι συναποφασίζουν ως προς αυτό το πρόγραμμα. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτόν τον λόγο είναι ε, απαραίτητο να λειτουργεί εύρυθμα. Και βέβαια εδώ υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες, υπάρχουν εθνικοί ε, και περιφερειακοί κανόνες που ισχύουν για τέτοιου ε, είδους ε, προγράμματος και βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζεται αντιμετωπίζει προβλήματα ε, το λέτε γιατί ε, πολλές φορές μόνο μία φορά η, ένα project ε, μπορεί να ε, υποστηριχθεί μόνο μία φορά από το πρόγραμμα και ακριβώς επειδή υπάρχει μόνο δυνατότητα μίας μόνο μοναδικής φοράς υποστήριξη και επειδή ακριβώς το κανονιστικό πλαίσιο είναι τόσο περίπλοκο υπάρχει μεγάλη δυσαρέστεια με αυτό και Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα ε, στο μέλλον. Ε, πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την Ευρώπη, αλλά το οποίο δυστυχώς συνοδεύεται από δυσαρέστια επειδή ε, διέπεται ακριβώς από ένα περίπλοκο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί και να μπορέσει να συμπορφωθεί με αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται με κάτι τέτοιο και δεν είναι επαγγελματίας σε αυτό το χώρο. Θεωρώ πως το Λίντερ έχει βελτιωθεί, αλλά υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης και νομίζω πως ε, σήμερα είναι σωστή χρονική συγκυρία για να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε από κοινού τι μπορούμε να βελτιώσουμε σε σχέση με το Leader μέσα στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να δούμε πώς μπορούμε να αντλήσουμε ακόμα περισσότερη προστιθέμενη αξία ε, και πώς μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα επιτόπου μέσω αυτού του προγράμματος. Επίσης, Υπάρχουν, βλέπουμε, και πολλές άλλες περιφέρειες και κοινότητες οι οποίες καταφέρνουν να χρηματοδοτήσουν πολλά περισσότερα μέσα του Λίντερ από ό,τι άλλα προγράμματα. Στο δικό μου το κρατήδιο, για παράδειγμα, τη Βάδη Βιτεβέργη, δεν έχουμε μόνο το κρατήδιο, αλλά έχουμε και 16 διαφορετικούς δήμους και κοινότητες και αν συγκρίνω το τι συμβαίνει για παράδειγμα στη Βαβαρία σε σύγκριση με αυτό που συμβαίνει στη Βάδη Βιτεβέργη, θα δω ότι στη Βαβαρία συμβαίνουν πολλά περισσότερα. Οπότε είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε σήμερα εδώ σε αυτή την ακρόαση μαζί μα ε, εκπροσώπους ακριβώς και από τι ε, ομάδε τοπική δράσης. Να ξεκινήσουμε όμως ε, κατευθείαν με την πρώτη παρουσίαση από την πλευρά τη κυρία Χόφμαν σε ό,τι αφορά του δείκτε αξιολόγηση των επιδόσεων στο πλαίσιο του Ρίντερ και βέβαια σα σας ευχαριστώ όλου και σας καλωσορίζω θερμά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Θα σας εξηγήσω καταρχήν το λιγότερο ίσως ελκυστικό για κάποιους τμήμα της πολιτικής που όμως είναι νευραλγικό τμήμα της πολιτικής, πολύ κρίσιμο. Αφορά τους δείκτες ελέγχου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Δηλαδή εξετάζεται η υλοποίηση, το αποτέλεσμα της πολιτικής και βλέπουμε πώς μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε, να το καταμετρήσουμε και να το ανακοινώσουμε. Καταρχήν να σας μιλήσω για τους δείκτες. Εδώ έχουμε κάπως ε, περίπλοκη ε, γραφική παράσταση. Ξεκινούμε από τους στόχους. Καταρχήν, τι είδους θέματα και στόχους ε, προωθεί το leader, σε τι μπορεί να συμβάλλει το leader. Και μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, βλέπουμε ποιοι είναι οι στόχοι της κοινή γεωργικής πολιτικής. Στη συνέχεια έχουμε πιο συγκεκριμένους στόχους για την αγροτική ανάπτυξη και βλέπουμε πώς το leader μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση αυτών των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης. Και από τους δείκτες υλοποίησης λαμβάνουμε άμεσες πληροφορίες για τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί. Αυτοί είναι οι δείκτες υλοποίησης και βλέπετε στο ροζ τετράγωνο τους δείκτες υλοποίησης που παρακολουθούμε, καταμετρούμε στα κράτη-μέλη και μετά τα κράτη-μέλη βάλουν εκθέσεις και έχουμε πολλές τέτοιες, τέτοιους δείκτες υλοποίησης όπως είναι οι δείκτες, το τμήμα πληθυσμό που αποκαλύπτεται από τις ομάδες τοπικής δράσης, το είδος των σχεδίων που χρηματοδοτείται από το Λίντερ και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια άμεσα ορατή πληροφορία για τους δείκτες υλοποίησης του leader. Επίση, συνδέουμε τις δράσεις με συγκεκριμένους στόχους. Εκεί καταμετρούμε τα αποτελέσματα που ε, διατίθενται σε αιτήσια βάση και εξετάζουμε δείκτες όπως το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από τις στρατηγικές, το ποσοστό του τοπικού πληθυσμού που καλύπτεται από τις βελτιωμένες υπηρεσίες και την υποδομή και βλέπουμε πόσες θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν χάρη στο Λίντερ. Και με τα αποτελέσματα αυτά και τις άμεσα αυτές συνέπειες των δραστηριοτήτων βλέπουμε πώς ε, πραγματοποιείται ο στόχος της αγροτικής ανάπτυξης που είναι η κοινωνική ένταξη, η μείωση της φτώχειας, η οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές ζώνες, γιατί θέλουμε να προωθήσουμε την τοπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές σε τελική ανάλυση. Και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να καταμετρήσουμε και τον αντίκτυπο. Να ευαθύνουμε δηλαδή στα αποτελέσματα του Λίντερ. Και εκεί έχουμε μία σειρά δικτών, όπως ε, το ποσοστό απασχόλησης, το κατακεφαλήνα ΕΠ, το συντελεστή, το ποσοστό φτώχειας. Και εκεί βλέπουμε ποια είναι η συμβολή ε, των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης γενικώ αυτούς τους δείκτες υλοποίησης, ε, δείκτες ε, αντικτύπου μάλλον. Αυτό είναι το σχέδιο, ο σκελετός αυτής της αξιολόγησης και μετά ε, περνάμε στην εφαρμογή. Ε, περνάμε σε ένα σύστημα καταμέτρησης αξιολόγησης πολιτικής με βάση τις επιδόσεις. Εδώ έχουμε δύο είδη δικτών που μας επιτρέπουν να εξετάσουμε την εφαρμογή. Δηλαδή καταμετρούμε την εφαρμογή σε αιτήσια βάση. Καταρχήν έχουμε τους δείκτες υλοποίησης και εδώ, για παρόμοια με τους δείκτες αυτής της περίοδου. Ε, προσδιορίζουμε τον αριθμό των δράσεων που έχουν δρομολογηθεί και βλέπουμε με τι δαπάνε σχετίζονται και τι προτείνει η, ε, η πολιτική για την ετήσια καθάριση απόδοσης προκειμένου να δοθεί αξιοπιστία για τις δαπάνες της ΚΑΠ, η δήλωση αξιοπιστίας. Δεύτερη κατηγορία δικτών στην παρακολούθηση και καταμέτρηση της εφαρμογής είναι δείκτες αποτελέσματος. Όπως είπα και προηγουμένως, συνδέουν μια δράση με, συγκεκριμένα, συγκεκριμένη πρόοδο. Δηλαδή τα κράτη-μέλη πρέπει να θέσουν κάποιους στόχους για αυτούς τους δείκτες αποτελέσματος και εμείς παρακολουθούμε την πρόοδο των προγραμμάτων βάσει αυτών των δικτών σε ετήσια βάση. Τώρα, σε μια πολυ... πολυετή προοπτική βρισκόμαστε στο μαύρο κουτί δεξιά με την, με την αξιολόγηση της πολιτικής, κάτι που γίνεται πιο μακροπρόθεσμα η πρόεδρος η κυρία Γκρέσλε είπε ότι μόνο μακροπρόθεσμα μπορεί κανείς να διαπιστώσει τα επιτεύγματα. Και αυτά τα καταματρούμε με δείκτες αντικτύπου που μας δείχνουν τις συνέπειες που είχαν για συγκεκριμένες πολιτικές στο Λίντερ και διάφορες παρεμβάσεις μας. Και στο νέο πλαίσιο μετά το 2020 θα σας παρουσιάσω τις πληροφορίες που θα έχουμε για το Leader, για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Leader, τι είδου δείκτες θα χρησιμοποιήσουμε εκεί για μετά το 2020 και πρώτα απ' όλα οι άμεσες πληροφορίε που δίνονται σε αιτήσια βάση για το Leader είναι ο αριθμό των τοπικών στρατηγικών που ισχύουν και που οι ομάδες τοπικής δράσης εφαρμόζουν επί τόπου. Και το χρησιμοποιούμε για την ετήσια μας ανάλυση. Αυτέ βέβαια οι στρατηγικέ μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη πολλών αποτελεσμάτων και οι πιθανές συνεισφορέ μπορούν να γίνουν ανάλογα με τη στρατηγική, τη φύση τη στρατηγικής και τι αποφασίζει ο τοπικός πληθυσμός να κάνει και μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Έχουμε δείκτες αποτελεσμάτων για τις νέε θέσει εργασία, δείκτε αποτελεσμάτων για τον τοπικό πληθυσμό που καλύπτονται από τη στρατηγική των έξυπνων χωριών και εκεί μπορεί να συμβάλλει το Leader. Επίσης έχουμε τον τοπικό πληθυσμό που επωφελείται από βελτιωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές. Έχουμε επίσης συγκεκριμένες ομάδες, ευάλωτες, μειονότητες που επωφελούνται από προγράμματα κοινωνικής στήριξης και κοινωνικής ένταξης και επίσης έχουμε ανάπτυξη επιχειρήσεων βιοοικονομίας. Αυτά τα παρακολουθούμε σε αιτήσια βάση και ενημερώμαστε για το τι συμβαίνει επί τόπου μέσω του Leader και τι αποτελέσματα αποφέρει το Leader. Τώρα, πιο μέσο και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εξετάσουμε τον αντίκτυπο του Leader για να δούμε σε τι βαθμό βοηθά το Λίντερ στην πρόθεση της απασχόλησης, στην κοινωνική ένταξη και την κοινωνική ανάπτυξη στις αγροτικές ζώνες, γιατί αυτός είναι ένα συγκεκριμένο στόχος της ΚΑΠ. Και εκεί χρησιμοποιούμε πληροφορίες για να καταμετρήσουμε την εξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης, του κατακεφαλήν ΑΕΠ, τη μείωση της φτώχειας, το, τα ποσοστά του τοπικού πληθυσμού και ούτω καθεξής. Είναι δείκτες που δεν προέρχονται από τα κράτη-μέλη, από τη Eurostat. Δηλαδή πρόκειται για γενικές πληροφορίες για την ανάπτυξη που παρατηρούμε στις αγροτικές περιοχές και που δείχνουν το βαθύτερο αντίκτυπο των μέτρων του Λίντερ. Μου ζητήσατε να σας μιλήσω και για τα ειδικά ιδιαίτερα επιτεύγματα του Leader. Τα πιο συγκεκριμένα επιτεύγματα του Leader. Θα σας δώσω καταρχήν ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να προσφέρει το Leader ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μας είπε και η κυρία Γκρέσλε για πολλά σημεία, το leader εφαρμόζεται τοπικά, περιφερειακά, είναι ένα πρόγραμμα και σχέδιο τοπικής ανάπτυξης, ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και ακριβώς ε, επειδή εκπορεύεται από την τοπική κοινωνία, έχουμε τερική σχέση συμμετοχική, χάρη στο leader και δημιουργούνται διάφοροι δεσμοί και διάφορες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων τομέων, κλάδων και εταίρων. Έχουμε οριζόντια και κατακόρυφη συνεργασία. Επίσης, καινοτομία είναι πολύ σημαντικό θέμα. Νέες αγορές, νέα προϊόντα αναπτύσσονται. Και ας μην ξεχνούμε και την κοινωνική καινοτομία που επίσης είναι πολύ σημαντική και πολύ σημαντικό επίσης θέμα. Ελοποιείται κάποια δικτύωση και ανταλλαγή των πρακτικών και κοινών λύσεων για κοινά προβλήματα. Αυτό προωθεί το Λίντερ μεταξύ άλλων. Και χάρη σε αυτή την εδαφική διάσταση και για πολλούς και άλλους λόγους το Λίντερ μας επιτρέπει να φέρουμε κοντά τους τον τοπικό πληθυσμό και μεταξύ του και με την Ευρώπη. Και αυτή είναι μια ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, να φέρουμε τον τοπικό πληθυσμό κοντά στην Ευρώπη. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά η κοινοί δείκτες που σας παρουσίασα είναι σχετικά εύκολα μετρήσιμη από τα κράτη-μέλη. Μια όμω και έχουμε πολύ διαφορετικές στρατηγικές επιτόπου. Οι, οι ιδιαίτερες ε, δυνατότητες του Λίντερ δεν καλύπτονται από τους γενικούς δείκτες, γιατί θα χρειαζόμασταν 100-150 δείκτες, γιατί το leader κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα ανάλογα με το πού εφαρμόζεται. Οπότε δίνεται διαφορετική έμφαση στην αξιολόγηση στα πλαίσια των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Και από αυτήν την άποψη, στην περίοδο 2014-2020, ζητήσαμε από τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης να, να κάνουν πολύ σοβαρές αναλύσεις, εδελεχείς αναλύσεις για το τι χρειαζόμαστε και προς τα που θα πρέπει να κατευθυνθούμε με ανάμειξη της τοπικής κοινότητας, των διαφόρων εταίρων, με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για να δούμε τι δράσεις θα αναλάβουμε. Επίσης, τοπικές κοινότητες θα πρέπει να ε, εντοπίζουν κάποιους ε, μετρήσιμους στόχους για την υλοποίηση και τα αποτελέσματα και να παρακολουθούν και να αξιολογούν όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Οπότε, οι ομάδες τοπικής δράσης υποχρεούνται να κάνουν αυτή την παρακολούθηση και την αξιολόγηση στα πλαίσια της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Και από εδώ προκύπτουν δύο δυνατότητες. Η μία είναι σε τοπικό επίπεδο, εκεί οι ομάδες τοπικής δράσης, LAGS λέγονται, χρησιμοποιούν την αξιολόγηση και την παρακολούθηση ως ε, εργαλείο διαχείρισης, βλέπουν ε, ποια είναι τα δυνατά σημεία, ποια είναι τα δύναμα που μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα και επίσης εξασφαλίζεται και ένας δημοκρατικός έλεγχος γιατί ο τοπικός πληθυσμός ε, βλέπει ποια είναι η έκβαση των δράσεων αυτών. Επίσης, οι ομάδες τοπικής δράσης δημιουργούν πληροφορίες και δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη μέσο και μακροπρόθεσμη αξιολόγηση. Έτσι δημιουργείται μια πολύ άρτια βάση για την αξιολόγηση του αντικτύπου του leader σε μεταγενέστερη φάση. Τώρα τι μπορεί να κάνει το leader, ποια είναι τα συγκεκριμένα του χαρακτηριστικά. Αυτά σας τα παρουσίασα και βλέπουμε κάποιους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων και αντικτύπου και υλοποίηση που καταμετρούν τα αποτελέσματα του leader. Βέβαια είναι ατελείς όλοι αυτοί οι δείκτες και ακριβώς είναι ευρύ το φάσμα των δραστηριοτήτων του leader και μεγάλες ε, ιδιαιτερότητες, γι' αυτό και δεν είναι πολύ ακριβείς όλοι οι δείκτες, αλλά θα πρέπει να βρούμε στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής ποια είναι η προστιθέμενη αξία του leader. Και βελτιώνοντας το κοινωνικό κεφάλαιο και δημιουργώντας ε, ικανότητες, διασυνδέσεις, επικοινωνία, εθελοντισμό. Στα πλαίσια της διακυβέρνησης έχουμε συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα πρώτα, πρότυπα μέτρα και δημιουργούμε έτσι πιο ανθεκτικές κοινότητες. Και αυτή η προστιθέμενη αξία θα πρέπει να εντοπιστεί, να καταμετρηθεί και να αξιολογηθεί επί τόπου στις, από τις ομάδες τοπικής δράσης της ΛΑΚΣ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα με τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Φιγκερέντο, που χθε παρουσίασε την γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου για την κοινή πολιτική. Τώρα θα μας μιλήσει για το ΛΙΝΤΕΡ και την προστιθέμενη αξία που έχει αυτό το πρόγραμμα. Γιατί δεν θέλουμε να ακούμε ότι τα δημόσια κονδύλια, τα κοινοτικά υποκαθιστούν τα εθνικά. Αλλά θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά όλα αυτά. Κύριε Φιγκερέντο, έχετε το λόγο. Πρώτα, πρώτα, λέει ο κύριος Φιγκερέντο, να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γεωργίας και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού γιατί κάλεσατε το Ελληνικό Συνέδριο. Θα σας ε, πω όσο γίνεται πιο σύντομα τη ισχύει για το Leader τι, ποια είναι η δική μας ε, αξιολόγηση. Να σας πω κάποιες ε, ιδέες για το leader σήμερα, αλλά επίσης και κάποιες άλλες σκέψεις για το μέλλον του leader εν ώψη της μεταρρύθμισης της ε, ΚΑΠ μετά το 2020. Με αυτή την προβολή PowerPoint θα δούμε που θα μας διευκολύνει το PowerPoint τι ισχύει. Πρώτα απ' όλα κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις δαπάνες. Το leader, κατά τη γνώμη μας, δεν ε, είναι ένας τομέας όπου δαπανούμε πάρα πολλά. Άρα δεν είχαμε το κίνητρο για να κάνουμε τον οικονομικό έλεγχο στο παρελθόν. Ε, αυτό πρώτα θα γίνει το 2010 και συνέχεια το 2012. Οπότε, αυτό θα πρέπει να εκτυπώσει το να ακούσετε τις ε, σκέψεις μας, ότι κατά κάποιο τρόπο τα συμπεράσματά μας ε, είναι λίγο ξεπερασμένα όσον αφορά όλους τους τομείς των δαπάνων και εάν Γόφερ πίνει η Επιτροπή Γεωργία ή Ελέγχου Προπολισμού θεωρεί ότι είναι σημαντικό το ελληνικό συνέδριο να ξανακάνει στο μέλλον οικονομικό έλεγχο, τότε μπορείτε να προκαλέσετε αυτή μας την ενέργεια, να το προτείνετε και εμείς ε, τα επόμενα χρόνια θα ε, το κάνουμε. Τώρα, τουλάχιστον 5% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη τη Υπέθρου θα πρέπει να πρεκοδοτήσει το Λίντερ. Υπάρχει ένας, ε, ένα ποσοστό χρηματοδότησης 20 με 80%. Και ήδη έχουν διατεθεί για το Λίντερ πάνω από 7 δις ευρώ. Μέχρι σήμερα πάντως ο ρυθμός απορρόφησης είναι χαμηλός ε, μόλις 11% από αυτά τα κονδύλια που έχουν διατεθεί. Ένα αυτό. Χαμηλό ποσοστό απορρόφησης. Τώρα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τα σχετικά με το leader, φαντασμό τα ξέρετε, αλλά θα πρέπει να το τονίσουμε και ξέρετε, εμένα μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Όπως ξέρετε, υπάρχει η μεθοδολογία από κάτω προς τα πάνω και με βάση την εταιρική σχέση και τη δημιουργία δικτύου. Αυτή είναι η μεθοδολογία όσον αφορά τις στατηγικές και είπαμε ότι καλύπτουμε 54% του πληθυσμού της υπαίθρου και το εφαρμόζουν ε, το πρόγραμμα, τέλο πάντων καλύτερα το πρόγραμμα, 2.745 τοπικέ ομάδε δράσης. Και πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι συμμετέχουν στο κόστος και στους κινδύνους. Υπάρχει μέσα αυτό το επιπλέον ε, στρώμα, το επιπλέον επίπεδο αυτών των τοπικών ε, ομάδων. Οπότε Έχουμε τώρα υψηλότερο κόστο και κινδύνου σε σχέση με τι παραδοσιακέ μεθόδου χρηματοδότηση. Αυτοί οι κίνδυνοι δικαιολογούνται από την προστιθέμενη αξία τέτοιων προγραμμάτων. Οπότε αυτό θα πρέπει να δούμε. Αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσουμε ακόμα και των προτέρων. Βλέπουμε τι προστιθέμενη αξία ε, επιτυγχάνεται με αυτό το πρόγραμμα. Και είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να αποδείξουν την ε, προσθέμενη αξία της προσέγγισης ε, αυτής για το λίτρο. Αυτό ήταν το συμπερασμά μας. Είπαμε ότι ήταν βέβαια δύσκολο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, γιατί υπήρχαν οι αγαθές προθέσεις, υπήρχε καλή πίστη και όπως σας είπα μου αρέσει εμένα αυτή η προσέγγιση, την έχω στην καρδιά μου. Όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι, αντικειμενικοί και θα πρέπει να μπορούμε να καταλήξουμε κάπου σε κάποιο συμπέρασμα. Τώρα, όσον αφορά το leader κατά την τρέχουσα περίοδο, θεωρούμε ότι επειδή υπάρχει ευξημένος κίνδυνος και δαπάνες, η εποπτεία και εξολόγηση του Λίντερ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στον αφορά την προστέμενη αξία. Έχουμε εδώ εννέα δείκτες. Εκτός από τους εθνικούς δείκτες. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι φορμοστικό χαρακτήρα. Δεν έχουν να κάνουμε τα αποτελέσματα γιατί μιλούμε για τις θέσεις απασχόλησης από τα έργα και σχέδια που καλύπτονται. Επομένω, βλέπετε ότι μόνο δύο δείκτες σχεδίζουν με αποτελέσματα, όλοι οι άλλοι δείκτες αφορούν την ε, υλοποίηση. Τώρα για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την παρακολούθηση κατά την τρέχουσα περίοδο. Έχουμε, είπαμε, πλέον τους εθνικούς δείκτες. Αυτό σε μια σειρά από περιοχές, σημεία στην Ευρώπη, για παράδειγμα στο Βέλγιο, συγκεκριμένα στη Φλάνδρα, υπάρχουν 8 με 10 δείκτες. με μια ματιά Περισσότεροι εξ αυτών έχουν να κάνουν με την υλοποίηση των ε, σχεδίων. Και μόνο μερικοί αφορούν τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση αυτή του Βελγίου έχουμε έναν για αποτελέσματα, έναν δίκτυο για αποτελέσματα και αφορά τα μεγαβάτη της ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία κάθε χρόνο μέσω του έργου παράγεται. Αυτό σαφώς ε, είναι ένα αποτέλεσμα. Όλοι οι άλλοι αφορούν κατάρτιση, εκτάρια. Λοιπόν, έχουν σχέση με την υλοποίηση, με την εφαρμογή του leader. Δεν αφορούν τα αποτελέσματά του. Όπως σας είπα, αυτοί οι δείκτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν την εφαρμογή υλοποίηση. Και στην προηγούμενη μας ε, ειδική έκθεση για το ΛΙΝΤΕΡ είπαμε ότι δεν υπάρχουν ε, ε, δείκτες αξιολόγησης και υπάρχουν πάρα πολύ λίγα επιστημονικά στοιχεία. Τα περισσότερα είναι συναισθηματικού επίπεδου, ούτως πεινεντυπώσεις. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες, περισσότεροι δείκτες όσον αφορά την υποστημένη αξία. Και ακριβώς ε, μια που υπάρχει ε, αυτό το πρόγραμμα με τέτοια κλίμακα και ποικιλία, του χρειάζονται διαφορετικές ε, προσεγγίσεις. Και σε αυτή την ειδική έκθεση διατυπώσαμε μια σειρά από συστάσεις. Τότε, 2012, είχαμε την συνέχεια και είπαμε ότι τα περισσότερα από αυτά είναι αποδεκτά και θα πρέπει να υλοποιηθούν. Άρα δηλαδή υπήρξε η τάση για καλύτερη αξιολόγηση. Τώρα στον πρώτο μέλλον της ε, ΚΑΠ το Λίντερ θα μοιάζει πολύ με το σημερινό. Αν κανείς μελετήσει τους προδυνόμενους κανονισμούς και τουλάχιστον 5% του Γεωργικού Ταμείου Ανάπτυξης Πέτρων θα καλύψει το Λίντερ και θα υπάρχει επίσης ποσοστό χρηματοδότηση που θα κυμαίνεται από το 20 μέχρι το 80%. Όμως η κοινωτική χρηματοδότηση θα εξαρτάται από τις επιλογές των κρατών μελών στα πλαίσια των στρατηγικών σχεδίων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Εμείς από πλευράς ελέγχου τονίζουμε αυτό το οποίο προείπαμε. Για όλα τα προτινόμενα όσον αφορά την αξιολόγηση. Δηλαδή θέλουμε ένα καλύτερο σύστημα επίδοσης το οποίο να επινοηθεί. Και όταν λέμε καλύτερη επίδοση, καλύτερο σύστημα αξιολόγησής της, εννοούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο συγκεκριμένοι πιο ποσοτικά αποτιμούμενοι στόχοι. Γιατί αν δεν είναι μετρήσιμοι, ε, αν δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν γίνεται. Άρα θα πρέπει να υπάρχει σαφή σχέση μεταξύ των δικτών και των ε, στόχων. Σε συνέχεια των όσων είπε η προλαλήσασα, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους κανονισμούς και έχουμε μόνο έναν δείκτη που τα προβλέπεται για το leader είναι η της τοπικής ανάπτυξης. Είναι ο στόχος 27 και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο δείκτης αλλά αφορά την υλοποίηση, αφορά την επίδοση. Είναι απλώς ο αριθμός των σχεδίων. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτός που θα εφαρμοστεί σε όλες τις αδικίες ή μόνο σε εκείνες που αφορούν την ε, υλοποίηση και εφαρμογή. Τώρα τι γίνεται με το 2020, ποια είναι τα συμπεράσματά μας όσον αφορά την αξιολόγηση στο μέλλον. Θεωρούμε ότι είναι περίπλοκο μέτρο το Λίντερ και η προσθέμενη αξία του σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό είναι κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο να αποτιμηθεί. Από τη μία μεριά η αποτίμηση κάποιων ε, πτυχών όπως η καινοτομία, η συνεργασία, το κοινωνικό κεφάλαιο, η δική διακυβέρνηση, όλα αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες στην αποτίμησή του. Από την άλλη μεριά θεωρούμε ότι οι σημερινοί προτινόμενοι δείκτες είναι μινιμαλιστική, είναι το ελάχιστο και απέχουν πολύ από το να μπορέσουν να συλλάβουν όλη την ε, ποικιλιομορφία του leader και της προσέγγισης του και την ε, ποικιλία επίσης των δυνατών δράσεων. Επομένω, χρειάζονται καινούργιοι δείκτες για να μπορέσουν να καλυφθούν όλες οι διαστάσεις, όλες οι πτυχέ του Λίντερ. Σα ευχαριστώ. Ναι, ε, αυτά που μας είπατε πραγματικά καταδεικνύουν όλα τα προβλήματα ακόμα περισσότερο και τώρα θα περάσουμε στον Άλιστερ Πράιορ από την σκοτσερική κυβέρνηση και τον επικεφαλή του ε, της ομάδας υποστήριξης ε, του περιφερειακού δικτύου. Σας ε, καλωσορίζουμε λοιπόν θερμά εδώ κύριε Πράιορ. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ μαζί μας και έχετε το λόγο. Um, thank you, Chair, for this opportunity to speak to you today about the implementation of the leader approach. Σε ευχαριστούμε που καλέσατε σήμερα εδώ να σας ε, παρουσιάσω τον αντίκτυπο ε, του Leader ε, στην δική μας κοινότητα αναφέρασε στον τίτλο της ακρόασης το Global Impact αλλά εγώ θα εστιάσω στη δική μου περίπτωση ειδικότερα από το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα από το 2007 και μετά. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, το πρόγραμμα 2007-2013, η προσέγγιση ε, LEADER εφαρμόστηκε από τη δική μας πλευρά με επένδυση 70 εκατομμύρια Βρετανικών λιρών. Και οι τοπικές στρατηγικέ ανάπτυξης ξεκίνησαν το 2008 με τα περισσότερα προγράμματα να έχουν καταστεί λειτουργικά από το 2012. Εγώ ήμουν υπεύθυνο ε, και για τα δύο προγράμματα Leader από την πλευρά τη κοτσική ε, κυβέρνηση από τι αρχέ του 2011 και ήταν σαφέ ότι είχαν αρχίσει να παρουσιάζονται κάποιε δογμέ, αν θέλετε, στο πρόγραμμα Leader, στο πρόγραμμα του προγράμματο αγροτική ανάπτυξη. Δηλαδή προβλήματα σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση από την πλευρά τη κυβέρνηση του Leader και το πώς αυτός ανήκε ή ήταν ολοκληρωμένο μέσα στα διαφορετικά ταμεία. Αυτές λοιπόν οι ρογμές, αυτά τα προβλήματα διαφάνηκαν ακόμα περισσότερο κατά το 2012-2013 καθώς ε, εκεί το καθεστώς των επιθεωρήσεων έγινε πιο αυστηρό και έγινε μια σειρά από επιθεωρήσεις. Εκεί λοιπόν αναγνωρίστηκαν μια σειρά από αδυναμίες σε όλα τα επίπεδα του προγράμματος. Και για μένα αυτό ε, πραγματικά μου δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό. Ε, καθώ υπήρχαν εκατοντάδε άτομα τα οποία αξιοποιούσαν το Λίντερ για να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή στην τοπική του ε, κοινότητα. Ε, μάλιστα, ένα, ε, υπήρξε μια πρωτοβουλία συνεργασίας για την διαχείριση των υδάτων διακοινωτικό μεταξύ δηλαδή Βρετανικής και Σκοτσαζικής κοινότητας και το οποίο πραγματικά έδωσε κίνητρα στους γεωργούς που συμμετείχαν να προέρχονται και σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και πραγματικά ε, αυτή το επιχειρηματικό πνεύμα που είχαν και η διάθεσή τους να επενδύσουν σε νέες συνδέσεις ήταν πραγματικά κάτι που με ε, εντυπωσίασε. Για την περίοδο 2007 έως 2013 εντοπίσαμε μια σειρά από προβλήματα στο Λίτερ. Δηλαδή, ε, συνολικά θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίθηκε στους στόχους του. Ναι, μάλλον δεν ανταποκρίθηκε. Το προσεγγίσαμε ενδεχομένως με λαθασμένο τρόπο εμεί το leader, ναι. Ίσως είχαμε μια λαθασμένη σκοπιά, ε, ναι. Και αν εγώ προσωπικά ήμουν δυσαρεστημένο, σίγουρα ε, ήμουν δυσαρεστημένο και ε, αντλήσαμε πολλά διδάγματα από αυτή την περίοδο του 2007 έως 2013. Περνάω λοιπόν τώρα στο Leader 2014 έως 2020 το οποίο αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαιρία για να ξεκινήσουμε πάλι εκ νέου και συμμετείχαμε σε μια σειρά από ε, workshops ε, αλλά και ε, μέσω του σημείου επαφή μα IRD, ώστε να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα Leaders στη Σκοτία. Και το σημείο αφετηρίας ήταν απλό. Θέλαμε να απλουστεύσουμε τη διαδικασία και να επιτρέψουμε στις εταιρικέ σχέσει να εφαρμόσουν τις στρατηγικές τοπική ανάπτυξη με τον τρόπο που εκείνες επιθυμούν και όχι με τον τρόπο που εμεί από την πλευρά τη διοίκηση επιθυμούμε. Φυσικά εντό πολύ συγκεκριμένων παραμέτρων. Και ε, είχαμε τις ομάδες ε, τοπικής δράσης οι οποίες εστίασαν ακριβώς στη στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης ε, έτσι ώστε να έχουμε τη σωστή προσέγγιση για να έρθει πραγματικά να λάβει ζωή, να λάβει σάρκα και οστά τον leader την περίοδο 2014-2020. Και φτάσαμε αντί για 33 μόνο σε 21 στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης. 14 από τις οποίες ήταν συγχρηματοδοτούμενες και από το EMFF και από το EFRT. Ε, και ε, με συνολικά 18-19 ε, εκατομμύρια λίρες που επενδύθηκαν σε τέτοιου είδους προγράμματα. Η FRD δηλαδή και η FF. και ποια ήταν η δική μας προσέγγιση. Καταρχήν είχαμε μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον, την κατανομή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τα εδάφη, την, τον πληθυσμό, αλλά και το, κοινωνικό-οικονομικό προφίλ της ε, κάθε περιοχής. Είχαμε επίσης ένα προϋπολογισμό 2 εκατομμύριο ε, ευρώ, ώστε να ε, έχουμε την κατάλληλη διοικητική διαχείριση. Και επίσης σε επίπεδο της καθοδήγησης μειώθηκε το σχετικό εγχειρίδιο κατά 100 σελίδες και φροντίσαμε να αναφέρουμε με σαφήνε τις προϋποθέσεις και δεν θέλαμε να είμαστε πολύ περιοριστικοί. Επίσης θέλαμε να έχουμε ένα πιο ελαφρύ κανονιστικό ε, πλαίσιο και επίση αναφερθήκαμε δηλαδή μόνο σε αυτό το πλαίσιο στις χρηματοδοτικούς κανόνες και στους κανόνες επιλεξιπότητες. Επίσης είχαμε ένα νέο σύστημα μηχανοργάνωσης ε, και επίσης ένα ε, δίκτυο συνεργασία. Και τώρα τι καταφέραμε από όλα αυτά. Καταρχήν επιτύχαμε μια πολύ πιο διαφανή διακυβέρνηση, δηλαδή έχουμε μια συγκεκριμένη ομάδα για την τοπική στρατηγική ανάπτυξη, έχουμε ένα ένα board, δηλαδή ένα συμβούλιο σε ό,τι αφορά ακριβώς την ανέλυψη της ευθύνης και έχουμε ένα δίκτυο προσωπικού LAG που λαμβάνουν υποστήριξη και αυτό το δίκτυο και το board από το ε, σκοτσέζικο δίκτυο. Επίσης έχουμε ένα πιο ισχυρό πλαίσιο τώρα, δηλαδή από, τις, από τους 250 και παραπάνω δείκτες εντοπίσαμε 30 δείκτες οι οποίοι είναι ιδιαίτερη χρήσιμη σε ό,τι αφορά τις 21 στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης στην ε, Σκοτία και επίση συνεχίσαμε και την ε, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε τοπικό επίπεδο και τώρα αστιαζόμαστε στην ε, αξιολόγηση ε, του Λίντερ και των αποτελεσμάτων των στρατηγικών αγροτική ανάπτυξης. Βασιζόμενοι βέβαια και στην αξιολόγηση του CLLD από το Help Desk. Άρα λοιπόν και εδώ πάλι αξιοποιούμε την εμπειρία και τα μαθήματα και τις πρακτικές άλλων συναδέλφων σε άλλα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα υπάρξει ε, από ό,τι γνωρίζουμε και από την Επιτροπή, ένα, μια ανασκόπηση των τελευταίων 20 ετών του Λίντερ, του ώστε να βοηθηθούμε καλύτερα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση στο μέλλον. Τώρα, τι έχουμε επιτύχει. Έχουμε ένα πολύ ε, πιο ισχυρό αγροτικό δίκτυο με ένα προπολογισμό 4 εκατομμυρίων λερών και ένα, ε, λιρών και ένα, μια ομάδα η οποία ε, ασχολείται με αυτό το τομέα. Έχουμε επίση περισσότερη έμφαση στην ε, στρατηγική ε, αγροτική ανάπτυξη και εδώ το leader βέβαια αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο αυτή τη στρατηγική και ε, ε, μόλι την τελευταία εβδομάδα είχαμε μια κοινή συνάντηση με το Αγροτικό Κοινοβούλιο, όπω λέγεται, τη Σκωτία και το οποίο κατέδειξε πόσο μεγάλη είναι η προστιθέμενη αξία του networking, της δικτύωσης δηλαδή, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος του leader για την ε, ε, ζωή των αγροτικών κοινοτήτων στη Σκωτία. Ε, κλείνοντας λοιπόν και συνοψίζοντας, ε, να πω ότι ο στόχος μας είναι να μειωθεί περισσότερο το διοικητικό άχθος έτσι ώστε να έχουμε και μια καλύτερη εφαρμογή του Leader. Αλλά δύο ακόμα στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω σε ό,τι αφορά το μέλλον του Leader. Πρώτον, ε, το Κοινοβούλιο το Αγροτικό της περασμένης εβδομάδας ε, κατέδειξε ότι και μου υπενθύμησε ότι πραγματικά οι μπορούν να ανταποκριθούν, μπορούν να καινοτομήσουν, να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες και υπάρχει αυτή η τάση δηλαδή ε, του να έχουν νέες ιδέες κάποιες, τις οποίες ακόμα δεν έχει υπάρξει άλλη ιδέα και αυτό καταδείχθηκε και με τις καινοτομίες ε, όπως αναφέρθηκαν στο Αγροτικό Κοινοβούλιο και στο ότι δηλαδή τέτοιου είδους καινοτομίες οδηγούν στην διευκόλυνση της ζωής των ανθρώπων στις τοπικές κοινότητες και δεν γνωρίζω να υπάρχει άλλο τέτοιο εργαλείο το οποίο ε, να μπορεί να καλύπτει τόσα διαφορετικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα ε, περίθαλψη για περιπτώσεις γεωτικής άνοιας μέχρι και ε, ευρυζωνικό ε, διαδίκτυο και ένα σωρό άλλα. Άρα λοιπόν το Αγροτικό Κοινοβούλιο εστιάζει ειδικότερα στι τοπικέ αγροτικέ ε, κοινότητε ε, ε, με τη διάσταση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γνωρίζουμε πω υπάρχει και η πρωτοβουλία των έξυπνων χωριών, αλλά λαμβάνοντα και υπόψη τι αρχέ αστική και αγροτική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν για την περίοδο μετά το 2020 οι ηθήνοντε θα έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να ανανεώσουν το leader, ώστε να προωθήσουν περισσότερο και την κοινωνική ισότητα στο στις αγροτικές κοινότητες. Αυτά από την πλευρά μου και σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Πολύ ενδιαφέρον ε, γιατί μας ε, παρουσιάσετε μια τοπική εμπειρία από το Λίντερ. Ε, ε τώρα από το ΕΛΑΤΖ έχουμε ένα μόνιμο εκπρόσωπο από την Νότια Ευρώπη ε, ο οποίο παρευρίσκεται σήμερα εδώ και πραγματικά μου ζήτησε διακαώ να πάρει το λόγο για δύο μόνο λεπτά. Παρακαλώ λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε, κυρίε και κύριοι. Έρχομαι από μια βόρεια περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα ε, να σας πω ότι ως ε, Γενικός Γραμματέας της, της μόνιμης ομάδας εργασίας που δημιουργήθηκε από τα ε, Υπουργέ Γεωργίας των ε, χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ε, θα ήθελα να σα παρουσιάσω τη δική μας άποψη για το Λίντερ. Εμείς κρίνουμε ότι το Λίντερ είναι πολύ χρήσιμο, χρήσιμο εργαλείο πολιτικής, καταρχήν για την ανάπτυξη της δημοκρατίας στις αγροτικές περιοχές και είναι γιατί στα πλαίσια του ΥΠΑΡΤ ξεκινήσαμε με μέτρα που μοιάζουν με αυτά του Λίντερ. Και μάλιστα η πιστοποίηση των μέτρων Λίντερ στη Μακεδονία, λέει ο μιλητής, ε, έχει προχωρήσει και ήδη έχουν γίνει, έχει γίνει όλη η νομοθετική προεργασία και το πρόγραμμα θα αρχίσει αμέσως. Ε, άλλες χώρες έχουν μείνει λίγο πιο πίσω, υστερούν κάπως. Πάντως, από πολιτική άποψη, την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια υπουργική διάσκεψη των Υπουργών Γεωργίας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων Και αυτή ήταν μια ευκαιρία να διατρανωθεί η πολιτική μας βούληση υπέρ της ε, ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα το Λίντερ ήταν ένα από τα θέματα που απασχολεί τους Υπουργούς Γεωργίας. Απ' την άλλη, όπως είδαμε, από την τρέχουσα εφαρμογή ε, μέτρων που μοιάζουν αυτά του Λίντερ στα Δυτικά Βαλκάνια, είναι ότι το πάθος, ο ενθουσιασμός του τοπικού πληθυσμού για τα μέτρα του Λίντερ, ή μέτρα που μοιάζουν με αυτό το Λίντερ, είναι, έρχεται σε αντίθεση με την ε, δινή οικονομική κατάσταση που είναι κάπως ζωφερή. Και μια και έχω λίγα λεπτά να σας παροτρύνω να κοιτάξετε την ιστοσελίδα μας με τις δημοσιεύσεις μας, τις ε, αναλύσεις, τις αξιολογήσεις που κάναμε για να δείτε τι κάνουν τα Δυτικά Βαλκάνια ως προς το Λίντερ. Και όποια και είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον του Λίντερ θα σταθούμε στο πλευρό σας. Πάντως για μας η πολιτική αυτή είναι από τις πιο σημαντικές και τις πιο επιτυχημένες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία 30 ετία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που επιστήσατε την προσοχή μας σε αυτή την πολύ σημαντική περιοχή που είναι τα Δυτικά Βαλκάνια και να δώσω το λόγο στην Ομίγερη ξεκινώντας από τον κύριο Αντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αχ, δεν περίμενα να είμαι ο πρώτος. Ευχαριστώ τους καλεσμένους μας και τον τελευταίο ομιλητή για την δική του μαρτυρία. Και είναι σημαντικό γιατί οι τοπικές κοινότητες δίνουν το στίγμα και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε προλαλή για τον άμεσο σύνδεσμο του Λίντερ με τη δημοκρατία. Και, και σημειολογικά, όταν μιλούμε για το Λίντερ, μιλούμε για την ε, εμπλοκή των τοπικών παραγόντων και των τοπικών κοινοτήτων για την τοπική ανάπτυξη. Και από το 1991 που ιδρύθηκε το Λίντερ καλό θα ήταν να έχουμε και δείκτες ε, για τους συνδέσμους μεταξύ των ε, συμμετεχόντων στο Leader. Περάσαμε από μια ε, γεωργική σε μια βιομηχανική κοινωνία και τώρα είμαστε σε μια υπερα... υπερατομικιστική κοινωνία. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να θέσουμε κάποια ζητήματα ουσίας και να δούμε μήπως η πολιτική με την ευρεία έννοια, την έννοια δηλαδή και της ε, συμβίωσης ε, σε μία επικράτεια, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και άλλους δείκτες πέραν του κατακεφαλής εισοδήματος ή της οικονομικής ανάπτυξης. Γιατί έχουμε και άλλες προκλήσεις, την κλιματική, την ενεργειακή, την περιβαλλοντική, τη βιοπικιλότητα, την υγεία των ανθρώπων. Και στο πρόγραμμα Leader και είμαι ευτυχώ ή δυστυχώς ε, από αυτού που παρακολούθησαν ε, το Λίντερ από τα Σπάργανα Νάτο το 1991 και είδαμε την εξέλιξή του και πώς έχει αναβαθμιστεί σε πραγματικό κοινοτικό πρόγραμμα αλλά δυστυχώ ε, το τυπικό διαδικαστικό τμήμα έχει πάρει το προβάδισμα σε σχέση με το ουσιαστικό. Θα πρέπει να επανακατευθύνουμε το leader και να σταθούμε στην πεμπτουσία του και όχι στον τύπο και τη διαδικασία. Γιατί η εμπλοκή της τοπικής κοινότητας και αυτό το δημοκρατικό στοιχείο βρίσκεται στην καρδιά του leader και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να πορευθούμε Και αν πάρουμε τους παραδοσιακούς δείκτες, τους κλασικούς, βλέπουμε ότι δεν αρκούν. Θα πρέπει να γίνει μια πολιτική γεωπολιτική αναθεώρηση και να καταλήξουμε σε νέους δείκτες. Επίσης, το δημοσιονομικό σκέλος που το επισήμανε ο κ. Φιγκερέντο από το ελεκτικό συνέδριο. Είναι μικρός ο δημοσιονομικός αντίκτυπος ε, του Λίντερ. Θα πρέπει να αναδείξουμε την πραγματική του αξία. Και έχουμε, θα έχουμε τις νέες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής μείωση κατά 27% του Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και Σίγουρα θα πληγεί και η αγροτική ανάπτυξη και ο δεύτερος πυλώνας με τις ε, νέες προτάσεις. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι αν περιοριστεί το κονδύλιο του Λίντερ θα πρέπει να αναθεωρήσουμε ίσως το περιεχόμενο και, και τα σχέδια που θα χρηματοδοτήσει στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της δημόσιας ακρόασης, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το πρόγραμμα LEADER. Θεωρώ ότι η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στο γεγονός ε, ότι εκπορεύεται από τις τοπικές κοινότητες και μακριά από τους πολιτικούς κύκλους. Αυτό που με προβλημάτισε κάπως ήταν τα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου για την προστιθέμενη αξία και την αποτελεσματικότητα του Λίντερ. Δεν θα επανέλθω στη χθεσινή συζήτηση ε, για την ουσία των προγραμμάτων που αποφασίζεται από τους πολιτικούς και όχι από το ελεκτικό συνέδριο. Αλλά ρωτώ το ελεκτικό συνέδριο πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την προστιθέμενη αξία μέσω των στοιχείων που ε, δίνουν οι ομάδες τοπικής δράσης. Γιατί ένας ε, εξοπλισμός ε, που σώζει ανθρώπινες ζωές είναι ανεκτήμητος. Δεν μπορούμε να το καταμετρήσουμε με απλό αριθμητικό υπολογισμό. Δεν θα πρέπει να έχουμε μια ρηχή ανάλυση του, της απορρόφησης των κοντιλίων. Στη Ρωμανία έχουμε την πανόλη των χείρων και είπαμε στις τοπικές αρχές να κατασκευάσουν αποτεφρωτήρες. Αλλά παρόλο που δεν ήταν μεγάλη επένδυση, δεν έγινε γιατί δεν τη θεώρησαν άξια λόγου. Χρειάζονται κάποια χρήματα για αυτά τα σχέδια τοπικής εμβέλειας που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής στην Ήπεθρο και αποτρέπουν την απερίμωση των αγροτικών περιοχών. Μόνο έτσι θα μείνει ο γεωρικός πληθυσμός στην Ήπεθρο βελτιώνοντα τι υπηρεσίε και τι υποδομέ. Σε ό,τι αφορά την περίοδο παρακολούθηση, εγώ θα την παρέτεινα από την πενταετία που ισχύει σήμερα στη δεκαετία. Θα πρέπει να καταμετρούμε την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και επίσης, καλά αυτά που γίνονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει η παρακολούθηση και ο συντονισμό να γίνεται από μια ευρωπαϊκή αρχή, γιατί είναι πιο εύκολο να έχει κάποιο τη γενική επισκόπηση αυτών των προγραμμάτων. Επίση, θα πρέπει να αυξήσουμε και τη χρηματοδότηση του Leader. Ενώ μα λένε ότι δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε κάποια κονδύλια για τι υπηρεσίε. Κι όμω πρέπει να κάνουμε κάποιε προκαταβολέ και για τι υπηρεσίε. Αλλιώ θα περιορίσουμε αισθητά την απορρόφηση των κονδύλιων, την εκταμίευση και θα εμποδίζουμε τη βραχία λυσίδα προμηθειών. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να τελειώσουμε αυτό το θέμα σε τρία λεπτά. Κυρία Γκονέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ce programme, je remercie euh, également, Να ευχαριστήσουμε και όλους όσους έλαβαν τον λόγο, λέει κύριε Γκλόνεκ. Μας προσθέσαν την ανάλυση τους για το πρόγραμμα. Επίσης και την κυρία Γκρέσλερ που μας είπε για αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο έχει κεφαλαιόδη σημασία για τον κόσμο και αναμφίβολα υπάρχει μια αντιστοιχία σε σχέση με το ε, τι θα, τι, τι εκπροσωπεί, τι στήριξε και από τον προπολογισμό αυτό το πρόγραμμα και τι δουλειά γίνεται στην πράξη. Αυτά τα προγράμματα τα διαχειρίζονται τα, οι ομάδες τοπικής δράσης, η κοινωνία δηλαδή. Αλλά όχι μόνο. Ακριβώς όπως ε, τόνισε ο συνάδελφος Αντριο, Δηλαδή, αυτά τα προγράμματα συνδέουν τη δημοκρατία με την κοινωνία. Και στη Γαλλία από το 2014 έχουμε την περιβραγή διοίκηση που κάνει τη διαχείριση. Άρα, από τότε που έγινε αυτή η μεταβίβαση αρμοδιότητας, συμμετέχουν οι περιφερειακές αρχές στα του προγραμματισμού. Και έτσι συνδέθηκαν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής με τους ε, στόχους ε, αυτών των ε, τοπικών αρχών. Επομένως ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη, πάρα πολύ θετική αυτή η μεθοδολογία, αυτή η οργάνωση συνδέθηκε η διοίκηση με την κοινωνία και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε και να το υπενθυμίζουμε κάθε φορά που μιλούμε για την ε, πρικοδότηση. Δηλαδή 5% περίπου 15% της πρικοδότησης για όλη την κοινή αγροτική πολιτική. Και το Ταμείο ανάπτυξη της Υπέθρου θα υποστεί την επόμενη χρήση 27% περικοπές. Οπότε όπως μπορούν όλοι να διαβεβαιώσουν από οποιαδήποτε θέση, πρόκειται για πολύ σημαντικό ε, πρόγραμμα για τους Ευρωπαίους. Καθένας πέτα πρόγραμματα από τη δική του σκοπιά, κύριε Φιγκερέντο, είπατε για την ε, απορρόφηση που φτάνει μόλις το 11%. Ασχολούμαι με την περιφερειακή δίκηση στη Γαλλία και ασχολούμαι με το θέμα της απορρόφησης και τις πληρωμές και ευρωπαϊκά και στη Γαλλία. Είμαστε στο 40%. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα αυτά και απευθύνουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να έχουμε δηλαδή αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία. Πρέπει να κλείσετε, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε και θεωρώ ότι για το εν λόγω πρόγραμμα ε, βασίλευε κάποια μικρή σύγχυση και νομίζω ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την άποψη όλων των εμπλεκομένων στην Ευρώπη όσον αφορά την ε, πάρα πολύ μεγάλη σημασία ε, του προγράμματος για τους Ευρωπαίους. Άρα αυτό ήθελα να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχουμε αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία για το σημαντικό πρόγραμμα. Και επίσης έχω έρθει σε επαφή με πολλές ε, ομάδες τοπικής δράσης. Και αυτά μου το τονίζουν συνεχώς. Ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Κύριε Σράιερ είναι η επόμενη ομιλητρία. Eh, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τα όσα μας εξήγησατε σήμερα το πρωί. Έχουμε κάποιον από τις κάτω χώρες. Δεν υπάρχει άλλος συμπατριώτης εδώ. Πάντως έχω εκπλαγεί από αυτά που ακούω. Ε, τέσσερα χρόνια είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο. Πάντοτε έχω κάποιους που με επισκέπτονται και προέρχονται από χωριά της Ολλανδίας και πάντοτε με ρωτάνε το πώς μπορούν να καλυφθούν από τα κοινωτικά κονδύλια. Γιατί μου λένε ότι προσπαθούν αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ναι, με ενδιαφέρει το θέμα των ομάδων τοπικής δράσης. Γιατί ξέρετε, όλοι οι φορείς των γυναικών ενδιαφέρονται. Είναι θέμα θέσεων εργασίας και θέμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μικροεπιχειρήσεων. Τι να σας πω, με που είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό απορρόφησης. Σας είπα, ο κόσμος διψάει για πρόσβαση στο πρόγραμμα στα κονδύλια. Οπότε, αν δεν θα γίνει, ιδίω με τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ. Είμαστε σε ώρες κρίσιμες πριν τις εκλογές θέλω όταν πάω πίσω στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια να μπορώ να τους απαντήσω σε ερωτήσεις τους. Και πήγα ας πούμε στο, στο Μπέρχεν ένα χωριό, μιλήσαμε για τα σχέδια με τους ε, δικούντες εκεί και ακριβώς λένε ότι δεν έχουν πρόσβαση στον κοινωνικό προϋπολογισμό ο επόμενο ομιλητή, ο αξιότιμο συνάδελφο Χόισλινγκ από του Πρασίνου. Σα ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που έχουμε σήμερα να ακούσουμε αυτές τις παρουσιάσεις και πραγματικά διαπιστώνουμε ότι το Leader είναι από τα πλέον καινοτόμα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ότι αποτελεί δηλαδή μια ευκαιρία δικτύωσης διαφορετικών ε, φορέων. Οπότε τίθεται βέβαια εύκολα το, το ερώτημα του γιατί υπάρχει απορρόφηση μόνο 11% από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Και αν δεν γνωρίζετε ούτε κι εσείς ε, ε, κύριε Σράιερ κάτι παραπάνω, τότε πραγματικά δεν γνωρίζουμε πολλά ως προς το τι συμβαίνει. Και δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή leader όπου ο αριθμός των φορέων είναι χαμηλός γιατί βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει κίνδυνος εμ, όχι κίνδυνος, συγγνώμη, φόβος σε σχέση ακριβώς με αυτές τις πολύ περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες και την ανάληψη της ευθύνης και ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις που τίθενται κατά πόσο ε, όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή αν θα ε, ανήκαν καλύτερα σε κάποιο άλλο δηλαδή όλα αυτά γίνονται ε, πολύ περίπλοκα για του Δήμου και τι κοινότητε για του περιφερειακού εφορεί, Οπότε θα πρέπει να πλουστεύσουμε λίγο τα πράγματα. Ο συντονιστή Λίτερμαν μα είπε ακριβώ ε, ότι χρειάζεται το μισό χρόνο από αυτό που δαπανεί μόνο και μόνο για να δει ποια προγράμματα ταιριάζουν πού ε, και σε ποιο πρόγραμμα. Οπότε ε, δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι λυπηρό και δεν μπορεί να συνεχιστεί το να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο προορίζεται για τι αγροτικέ κοινότητε και το οποίο δεν αξιοποιείται τελικά σε μεγάλο βαθμό. Ε, δεν μπορεί δηλαδή να αποτελεί υπόδειγμα για άλλε περιοχέ, ακόμα και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αξιοποιείται. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, ε, και προτού δώσω το λόγο ε, στους εμπειρογνώμονες για να δώσουν πολύ σύντομες απαντήσεις. Να δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή από τους συναδέλφους του κύριο Φλανάκα. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του Λίντερ, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από το Λίντερ, όπου και αν κοιτάξω ε, στην ε, δική μου κομμόπολη. Ε, σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, δεν είχαμε για παράδειγμα κανέναν τομέα χώρο που θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε για παράδειγμα μια θεατρική παράσταση έχουμε ε, κάποια σημεία ε, ε, περιπάτων ή κάποιες διαδρομές καγιάκιν για παράδειγμα που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε με άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν με διάφορους τρόπους το Λίτερ πραγματικά κατάφερε να έχει μαζικό αντίκτυπο. Ναι, ίσως υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της επιτυχίας του Λίτερ αλλά σας λέω πραγματικά ότι όπου κι αν κοιτάξω υπάρχει επιτυχία, υπάρχει αποτέλεσμα από το Λίτερ. Ε, εκείνο τελικά που οδήγησε για παράδειγμα στην, στο, στη διακοπή του προγράμματο για το Καγιάκι είναι ακριβώ ο περίπλοκο ε, χαρακτήρα τη διαδικασία για να έχει κανεί ε, πρόσβαση στα κονδύλια. Δηλαδή τελικά ορισμένε περιπτώσει αναφέρθηκε ότι καλύτερο θα ήταν να έχουμε πάρει ένα δάνειο ώστε να μην χρειαστεί να υποβληθούμε σε όλη αυτή την περίπλοκη διαδικασία. Οπότε είναι λίγο ε, ηρωνικό το ζήτημα του ότι συζητάμε εδώ την αξία των κονδυλίων τα οποία αξιοποιούνται στο Λίντερ. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ε, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι αποφελούνται από το Λίντερ τη σήμερα ημέρα εργάζονται με βάση τα όσα κατάφεραν. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για τους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Πού είναι όλοι οι συνάδελφοι για μία ακόμα φορά σήμερα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Λόζικοφμα λοιπόν ως πρώτη για να δώσει απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Ε, ακούσαμε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες με το Leader, αλλά πολλές ε, τις διορθώσαμε με τη νέα νομοθεσία για την περίοδο αυτή. Και η ιδέα να έχουμε στο μέλλον μόνο ένα δίκτυο για το Leader δεν ισχύει. Έχουμε τουλάχιστον πέντε δείκτες αποτελεσμάτων ε, και τέσσερις αντικτύπου. Βέβαια έχουμε περιορισμένες ε, δυνατότητες ε, καταμέτρηση σε τόσο αφηρημένο επίπεδο. Και αυτό που φάνηκε από τους ε, ομιλητές καλεσμένους είναι ότι θα πρέπει να πάμε επιτόπου και να καταμετρήσουμε εκεί τα αποτελέσματα. Και αυτό κάνει και το νέο σύστημα που προτείνουμε. Να έχουμε μια αξιολόγηση της στρατηγικής επιτόπου για να καταλήξουμε σε πιο ειδικού δείκτες. Γιατί αν αυτό το κάνουμε σε κοινοτικό επίπεδο ευρωπαϊκό, ε, ερχόμαστε στην κατάσταση του σκοτσέζικου προγράμματος που έχει 250 μεμονωμένους δείκτες. Θα ήταν πολύ δύσκολο να το προβάλλουμε κάτι τέτοιο και να γίνει αποδεκτό από τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχει υποχρέωση υποβολή εκθέσεων για το Λίντερ. Θα πρέπει λοιπόν να καταβούμε σε τοπικό επίπεδο στη βάση με τοπικού δείκτε που θα είναι πιο προσαρμοσμένοι και πιο εκλεπτισμένοι. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δαπανών και τα προβλήματα με τις δαπάνες. Εμείς μέχρι στιγμής ε, για το Λίντερ έχουμε δώσει 14% του προϋπολογισμού. Είναι χαμηλό το ποσοστό, γιατί για την αγροτική ανάπτυξη έχουμε καταβάλει το 33%. Αλλά το Leader ε, ε, έχει πιο χρονοβόρες διαδικασίες για να ξεκινήσουν κάποια θέματα και Μακάρι να μπορούσαμε να τα επιταχύνουμε, αλλά η κατάσταση έτσι έχει. Πάντως, το 36% του προϋπολογισμού ήδη έχει δεσμευθεί για συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια και ειδικέ δράσεις για το θέμα αυτό, για το Leader. Και βέβαια έγινε μια καθυστερημένη έναρξη του Leader και σωστά επισημάθηκε γιατί είναι περίπλοκο το σύστημα του Λίντερ και απαιτούνται πολλά δικαιολογητικά για τις δαπάνες και για τις επιλογές που κάνουν τα κράτη-μέλη και οι ομάδες τοπικής δράσης. Κάτι που προποθέτει παροχή πληθώρας πληροφοριών, κάτι που δεν είναι εύκολο από τους ντόπιου να χορηγήσουν τόσε πολλές πληροφορίες. Επίσης, τα κράτη-μέλη ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση να εφαρμόζουν το Leader. Και μάλιστα είναι πολύ μεγάλο κράτος μέλος. Ε, μόνο το τελευταίο μήνα επέτρεψε την υποβολή αιτήσεων για το Leader. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να επεκτείνει τα συστήματα πληροφορίες και τεχνολογίες ε, για το Leader. Εξού και οι καθυστερήσεις. Ο κύριος Φιγκερέντε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Όπως είπε και στην αρχική μου ομιλία, η συμπάθεια προς τέτοιο είδους προσεγγίσεις είναι μεγάλη, αλλά το θέμα δεν είναι η συμπάθεια. Δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό, πόσο συμπαθούμε ή μας αρέσει ένα πρόγραμμα. Το πιο σημαντικό είναι οι δείκτες, γιατί πολλοί θα πούν «Α, το ελεκτικό συνέδριο μόνο προβλήματα μας δημιουργεί» ε, και εμποδίζει την ανάπτυξη των σχεδίων το ελεκτικό συνέδριο, παρεμποδίζει τις επενδύσεις. Όχι. Το θέμα δεν υπάρχει. Δεν, υπάρχει. δεν θέτει το ελεκτικό συνέδριο κανένα πρόβλημα στην εξέλιξη των σχεδίων. Αυτό που λέμε στο ελεκτικό συνέδριο είναι ότι θα πρέπει να μπορούμε να καταμετρούμε τα αποτελέσματα. Γιατί αν έχουμε αποτελέσματα καταμετρήσιμα θα είναι πολύ πιο εύκολο και σε πολιτικό επίπεδο να προωθήσουμε προγράμματα σαν το Leader. Γιατί θα έχουν αποδειχθεί τα αποτελέσματά τους. Και για μας το σημαντικό είναι οι δείκτες, οι δείκτες αποτελέσματος και όχι οι δείκτες εφαρμογής. Και όταν λέμε ότι θα πρέπει να παρατείνουμε την περίοδο των επενδύσεων και να την επεκτείνουμε στην δεκαετία, Θέλουμε να είναι πιο αποτελεσματικέ, λέτε, οι επενδύσει. Γι' αυτό θέλετε παράταση προθεσμία. Και πώ θα καταμετρήσουμε την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα των επενδύσεων. Κάπω θα πρέπει να το κάνουμε. Γιατί αν δεν έχουμε αξιόπιστου δείκτε, πώ θα αποδειχθεί αυτή η αποτελεσματικότητα ή η αποδοτικότητα. Θα πρέπει κάπω να αποδειχθεί. Αλλιώ είναι δύσκολο να αναπτύξουμε αυτά τα προγράμματα μικρή εμβέλεια μέσω του Λίντερ. Ευχαριστώ. Τέλος ο Συμφωνώ. Πολλά θετικά θα μπορούσαμε να πούμε για το Λίντερ όσον αφορά τις επιπτώσεις για τον κόσμο. Βέβαια, η γραφειοκρατία ανέκαθεν ήταν το πρόβλημα που επισημαίνουν οι πολίτες. θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Είναι το θέμα και η πληροφορική, δηλαδή πώς γίνεται η εφαρμογή από τις ε, τοπικές ομάδες δράσης, αλλά σε εκείνο το επίπεδο θα πρέπει να δούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, να βοηθήσουμε αυτές τις ε, ομάδες και τα πράγματα να μην μπερδεύονται περισσότερο από όσο χρειάζεται. Είπαμε ότι έχουμε 250 δείκτες στην Σκοτία. 21 στρατηγικές, ε, τόσοι πολλοί δείκτες είναι προς απορία. Και προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η συνολική εικόνα. Πρέπει να δούμε πώς βελτιώσουν τις στρατηγικές από τις ε, ομάδες τοπικής δράσης και να δούμε τελικά ποιοι είναι οι δείκτη που χρειάζονται για τις ανάγκες τους. Και πώς θα θέσαμε να βοηθήσουμε, το πώς θα γίνουν πιο ρεαλιστές, πώς θα χρησιμοποιήσουν πιο αφιώς το σύστημα. Αν κανείς θέλει να καταλάβει το leader, θα πρέπει να υπάρχει η σωστή προσέγγιση για την αξιολόγηση και βέβαια προς τούτο χρειάζονται οι κατάλληλοι δείκτες. Δεν είπα στην εισηγησή μου ότι η εμπειρία μας στη Σκοτία κατέδειξε ότι κάθε επένδυση αξίζει ότι όλα απορροφήθηκαν, όλα πιάσανε τόπο. Αν χρειάζονται. Ε, και αυτό δείχνει ότι ε, αξίζουν τα χρήματα που επενδύονται στο leader. Αυτό μπορεί να είναι για τη σημερινή συζήτηση. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα... Ε, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο της μέσα διάταξης και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Στο δεύτερο πάνελ. Έχω την ευχαρίστηση να το να αρχίσουμε τη ζήτηση τώρα και τώρα θα ασχοληθούμε με την τοπική πτυχή του θέματος και με τα, με, τα καινοτόμα του leader. Οπότε θεωρούμε ότι μπορούμε να εμβαθύνουμε και να βελτιώσουμε το λειτουργία το μέλλον. Και γι' αυτό έχουμε τώρα τους ειδικούς μας. Πρώτη η Μαρία Ζωμποτέλιο που είναι πρόεδρος του φορέα Leader για την ανάπτυξη της ε, Υπέδρου. Έρχεται από την Πορτογαλία. Πριν της δώσω το λόγο, υπενθυμίζω δεν έχετε 10 λεπτά. Έχετε 9,5 λεπτά, λέει ο πρόεδρο. Ε, começo por agradecer ao Comitê de Agricultura e Desenvolvimento Rural e ao Comitê do Controlo. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπέθρου και την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών για αυτήν την ε, πρόσκληση σήμερα εδώ και τη οργάνωση της ακρόασης. Η Ελλάδα που δημιουργήθηκε το 1999 ε, αντιπροσωπεύει 2.500 ε, ομάδες τοπική δράση από 25 ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 23 μάλλον κράτη-μέλη και δύο γειτονικά κράτη, το οποίο βέβαια καταδεικνύει και το ενδιαφέρον που υπάρχει για το Leader εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του ΕΛΑΡΤ είναι να προωθήσει μια ε, καλύτερη ποιότητα ζωής στις αγροτικές ε, περιοχέ μέσω τη παραμονή και των σχετικών ε, πληθυσμών σε αυτέ τι περιοχέ, αλλά και η διάδοση τη μεθοδολογία Leader και η ενίσχυση και η βελτίωση της, του μηχανισμού τη τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Και σήμερα θα κάνω μια παρουσίαση αυτών των τοπικών εταιρικών σχέσεων και θα κάνω και κάποιε κάποιες κάποιε προτάσει προτάσεις, θα αναφερθώ στις προκλήσεις μας. Ε, με βάση λοιπόν τη δική μας ανάλυση στην εξέλιξη του Λίντερ από το 1991 υπήρξαν δύο σημαντικά ορόσημα ε, τα οποία αποτέλεσαν ευκαιρίες οι οποίες όσο δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως. Καταρχήν η ενσωμάτωση του Λίντερ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στην ε, περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και Παραλαμβάνω λοιπόν δύο δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως. Αφενός οι οποίες η δυο οροσημα τα οποια δεν αξιοποιηθηκαν πληρω αφενος η ενσωματωση του Λίντερ στα προγράμματα ε, τη ανάπτυξης ανάπτυξη στην περίοδο 2007-2013 και ο πολυτάμιακος χαρακτήρας του μηχανισμού για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών ε, κοινοτήτων, ε, ο οποίος υιοθετήθηκε μόνο σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ο Λίντερ λοιπόν ε, αποτέλεσε μια πρωτοποριακή ε, πρωτοβουλία, ώστε να προωθήσει νέο είδου σχέση ανάμεσα στι δημόσιε αρχέ και την κοινωνία των πολιτών. Ε, Προωθώντα λοιπόν ένα νέο τρόπο διακυβέρνηση, όπου υπάρχουν διαφορετικοί φορεί οι οποίοι έχουν πλέον νομιμότητα για, και πρόσβαση στα δημόσια κονδύλια χρηματοδότηση και ε, δρούν από κοινού στο πλαίσιο του, του, <clears throat> της πολιτικής ζωής με περισσότερη αυτονομία Αυτή λοιπόν η ε, προσέγγιση ε, επέτρεψε μια ε, άμεση σχέση μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων με την ε, με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και ακόμα και αν δημιουργήθηκε μέσα στην κοινή γεωργική πολιτική, το Leader ε, έφερε τις επενδύσεις της Ευρώπης στις αγροτικές ζώνες και όχι μόνο στον τομέα της γεωργίας. Δηλαδή βοήθησε στον εκδημοκρατισμό της διαχείρισης ακριβώς μέσω της συμμετοχικής του μεθοδολογίας αλλά και συνέβαλε στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στα δημόσια κονδύλια. Κατά τα τελευταία 27 χρόνια το δίκτυο των ομάδων τοπικής δράσης συνέχισε ξανά και ε, καταδεικνύει και ότι υπάρχει και ενδιαφέρον για αυτόν τον νέο τρόπο διαχείρισης ε, ε, των της, ε, αυτής της ε, πολιτικής ε, γιατί ακριβώς έδωσε το παράδειγμα και σε άλλες χώρες όπως η Γεωργία, τη Μολδαβία, τη Μοζαβίκη και πιο πρόσφατα στην Κίνα. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις μεταβατικές περιόδους ανάμεσα στις περιόδους προγραμματισμού αναφέρονται ξανά και ξανά αμφιβολία σε ό,τι αφορά την προστέμενη αξία του leader. Και βλέπουμε ότι στα δεδομένα ε, παρακολούθησης των ε, προγραμμάτων ε, αγροτικής ανάπτυξης να υπάρχει γενικότερα χαμηλή συμμετοχή και χαμηλός βαθμός υλοποίησης των μέτρων leaders σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, το οποίο βέβαια αποτελεί λογική συνέπεια της καθυστέρησης σε ό,τι αφορά τις προσκλήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή των ομάδων τοπικής δράσης. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζουμε την νέα δημοσιονομική πρόταση για την περίοδο μετά το 2020 που μειώνει ε, σε ένα έτος, στην περίοδο των δύο ετών σε ό,τι αφορά την ε, έγκριση των ομάδων τοπικής δράσης. Γιατί αυτό θα επιτρέψει ακριβώς το να μειωθούν, να κλείσουν αυτά τα κενά που υπάρχουν στις μεταβατικές περιόδους. Ε, ε, αν θέλουμε να έχουμε να αξιολόγηση μια δημόσια πολιτική, τότε θα πρέπει να αξιολογήσουμε τη λογική τη, του στόχου τη και ότι ακριβώ θέλει να επιτύχει τι δηλαδή προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτό το λίγο, τι προσπάθησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1991 και σε ποιο βαθμό αξιοποιήθηκαν τα σχετικά εργαλεία. που οδηγούν στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι στο, κατά τον τερματισμό της ε, ε τρέχουσας ε, περίοδος ε, προγραμματισμού ε, έχουμε το, σύστημα, το κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης και εκεί βέβαια θα βρούμε ε, ως δείκτε μόνο για παράδειγμα των ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται και τη δημιουργία των θέσεων εργασία, Αλλά αυτό δεν επαρκεί. δεν μπορούμε δηλαδή, δεν μετρούμε το κοινωνικό καφέλο το οποίο δημιουργείται, τι νέε πρακτικέ οι οποίες ε, ε, ε, επιτυχάνονται, αλλά και την αλλαγή τη νοοτροπία, η οποία λαμβάνει η χώρα. ακόμα και η, η εμβάθυνση αν θέλετε των ταυτοτήτων στις αγροτικές κοινοτήτες με περισσότερες πρωτοβουλίες, με ε, περισσότερες υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν λόγω ακριβώς του τοπικού χαρακτήρα των ομάδων τοπικής δράση και λόγω του πολυτομιακού ε, ε, χαρακτήρα υπάρχει ε, δυσκολία στο να μετρηθούν ακριβώς με απτό χαρακτήρα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουν τα μέτρα του Λίντερ. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να τίθεται ένα αμφιβόλο η προστέμενη αξία του Λίντερ. Ο νομοθετικό πακέτο που προτάθηκε από την Επιτροπή στα τέλη του Μαΐου ε, σε ορισμένο ε, βαθμό περιορίζει τις δικές μας φιλοδοξίες ε, και γι' αυτό προσπαθούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας εδώ ώστε να υπάρξει αναθεώρηση. Θεωρούμε δηλαδή λοιπόν το γεγονός ότι το ΦΕΝΤΕΡ δεν ανήκει πλέον στα ε, και επενδυτικά ταμεία και γιατί θεωρούμε πως αυτό αποτελεί οπισθοχώρηση και τελικά για όσους συμμετέχουν στις ομάδες τοπικής δράσης δυσκολεύουν τα πράγματα. Η δυνατότητα λοιπόν των, της των ε, ε σχετικών κανόνων ε, του, γενικού, του, του, του, βασικού ταμείου είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή θεωρούμε πως είναι εσφαλμένο ε, να διαχωρίσουμε την ε, αγροτική ε, ανάπτυξη από την πολιτική συνοχή. Γιατί ακριβώ αυτή η αγροτική ανάπτυξη έχει και μια πολύ σημαντική κοινωνική διάσταση, αφού έχει και άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωή των αγροτικών κοινοτήτων. Άρα λοιπόν η διαδικασία, ε, η διευκόλυνση τη πρόσβαση τη διαχείριση και η εναρμόνιση των σχετικών διαδικασιών σε ό,τι αφορά τα ταμεία είναι πάρα πολύ σημαντική αν ακολουθήσουμε αυτή την ε, λογική, τότε η αγροτική διάσταση ε, του ΦΕΔ μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ε, και δεν θα βγει τελικά περισσότερο αποδυναμωμένο για το Λίντερ. Και εδώ χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενισχύσει τον προπολογισμό της Ένωσης μέσω του νέου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθεί μια πολιτική συνοχή αλλά και μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική. Ε, και ε, επίσης θεωρούμε ότι σε αυτές οι δύο σημαντικές πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να ε, προετοιμάζονται και να εφαρμόζονται με πιο συντονισμένο τρόπο και προωθώντας περισσότερο τις συνέργειες. Οι δύο τελευταίες εκδοχές του Leader και το εργαλείο του CLLD μπορούν να μας δώσουν κάποια διδάγματα, μπορούν να μας δείξουν πώς μπορούν να αποφύγουμε τα ίδια ασφάλματα στο μέλλον. Ε, θα πρέπει για παράδειγμα να αντιμετωπίσουμε την πολυπλοκότητα των ε, ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές ε, κοινότητες με αντίστοιχο τρόπο, όχι δηλαδή με, ένα πολύ περιορισμένη, με πολύ περιορισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά μόνο το δεύτερο πυλώνα τη κοινωνική πολιτική και το αφέντερ. Και επίση, αν θέλουμε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη, θα πρέπει να καλύψουμε διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κονδύλια από διαφορετικά ταμεία. Η εφαρμογή ταυτόχρονα ε, του CLLD ε, καθιστά απαραίτητα μια, ένα πολύ καλό συντονισμό ανάμεσα σε διάφορες αρμόδιε διαχειριστικέ αρχέ, αυτό που δεν έχει δηλαδή συμβεί μέχρι στιγμή. Ε, Επίση, οι περιορισμοί στον προπολογισμό και το διοικητικό άχθο, και μάλιστα υπερβολικό διοικητικό ε, περιορίζουν τι δυνατότητε που έχουν οι ομάδες τοπική δράσης ώστε να προωθήσουν την αγροτική ανάπτυξη. Ε, άρα λοιπόν χρειάζεται ε, να γίνει αυξημένη χρήση των δυνατοτήτων απλουστευμένων ταπανών και η περισσότερη απλούστευση των ίδιων των διαδικασιών. θα πρέπει δηλαδή οι ομάδε τοπική δράση να θεωρηθούν ω φορεί οι οποίοι συναποφασίζουν σε ό,τι αφορά την πολιτική αγροτική ανάπτυξη και έχουν τη δική του ταυτότητα. Γιατί αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ανοικοδόμησή τη είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που θα πρέπει να επιτύχει το Λίντερ. Σε επίπεδο ε, ευρωπαϊκό τώρα η Έλλαρντ έχει παρακολουθήσει ε, όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει και ε, στα τέλη του προηγούμενου έτους συντάξαμε ένα έγγραφο σε ό,τι ακριβώς αφορά την ανανέωση του Λίντερ και της CLLD και διαβιβάσαμε αυτή την, αυτό το έγγραφό μα ε, στι κυβερνήσει των κρατών μελών. Σε αυτό λοιπόν μα το έγγραφο, σε αυτό το μοντέλο, τι υπερασπιζόμαστε, την ε, απλούστευση του leader ε, ε, καθόλου σε όλα τα στάδια τη υλοποίηση, η δημιουργία ενό αποθεματικού ταμείου στο οποίο θα συνεισφέρουν όλα τα επενδυτικά και τα αθωτικά ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενό επιχειρησιακού προγράμματο leader CLD σε κάθε κράτο μέλο. Ε, με συγκεκριμένους κοινού απλού κανόνε, όπω έχει ήδη δημιουργηθεί για παράδειγμα στην ε, Σουηδία. Ε, και επίση υποστηρίζουμε ότι ε, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχουν όλε τι δυνατότητε επιλογή τη ομάδα τοπική δράση ό,τι αφορά τα μέτρα που θέλουν να υλοποιήσουν και δεν θα πρέπει το Λίντερ να αποτελεί ένα μενού από το οποίο δηλαδή στο οποίο προσθέτουν ό,τι θέλουν οι αρμόδιε κυβερνήσει. Στο τέλος του, στα τέλη του Σεπτεμβρίου η Ελλάδα προέβη στην διοργάνωση μια εκδήλωση όπου συμμετείχαν 300 εκπρόσωποι από 27 διαφορετικά κράτη-μέλη. Και αναφερθήκαμε λοιπόν πολύ σε προβλήματα τα οποία έχουν πολυτομιακό χαρακτήρα. Άρα λοιπόν στο ε, πλαίσιο της μείωσης του προπολογισμού για την κοινή και οργική πολιτική, ε, όπου προβλέπεται μόνο το 5% του Φέντερ για το Λίντερ και αρμοδιότητα λήψη αποφάσεων και πάλι για τα κράτη-μέλη, υπάρχει ο κίνδυνο, ε, τα κράτη-μέλη να μην αξιοποιήσουν ούτε καν αυτό το 5%. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή θα έπρεπε να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να μην περιοριστεί μόνο στο 5% και από την άλλη πλευρά να επαληθεύει ότι εφαρμόζει τη μεθοδολογία ε, του Λίντερ. Άρα λοιπόν προτείνουμε το από 5% σε 10% να πάει το ε, ελάχιστο ποσοστό η ελάχιστη, το ελάχιστο ποσοστό του Φέντερ για το Λίτερ και ε, τουλάχιστον 80% συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες αυτά τα μέτρα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σε αυτό το πλαίσιο και αξιοποίηση της τοπικής εμπειρίας αλλά και ευέλικτο συνδυασμό των ευρωπαϊκών, των ενωσιακών δηλαδή κοντιλίων αλλά και των εθνικών και ατομικών ε, κονδυλίων. Ε, θεωρούμε πως και είμαστε πεπισμένοι ότι με τα 25 χρόνια ήδη εργασία που έχουν πίσω του οι ομάδε τοπική ανάπτυξη μπορούν να συμβάλλουν πραγματικά στο να διατηρηθούν ζωντανέ ε, τα εδάφη και οι κοινότητε περιφερειακέ τη Ευρώπη. Οι ε, προκλήσει λοιπόν που αντιμετωπίζουν μα ε, αναγκάζουν να είμαστε να επαγνωγούν πιο πολύ και να μην επιτρέπουμε το να υποτιμούνται τέτοιου είδους τομεακές πολιτικές η συμμετοχή λοιπόν των τοπικών φορέων ε, στον καθορισμό των προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις αλλά και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των πολιτικών ε, ε, μέτρων είναι ζωτική σημασία ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα να υπάρχει καλύτερη σχέση κόστος αποτελέσματος αλλά και περισσότερη εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λαμβάνοντα υπόψη τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση και του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, θεωρούμε πω οι ομάδε τοπική δράση μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εδαφών, ε, βρίσκοντα λύσει ε, ε, για τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι κοινότητε, λύσει οι οποίε μπορούν να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο συνεκτική και πιο αλληλέγγυη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για όσα μα είπατε, για όσα μα προτείνατε, κύριε Μποτέλη. Και τώρα έχουμε τον κύριο Ρικάρντο Φαρτζόνη. Έχετε 10 λεπτά, κύριε. Eh, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, εξαιρετικοί κύριοι βουλευτές. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα δέκα λεπτά που μου διαθέσατε και θα πρέπει να σα ε, πω σύντομα τι ισχύει και να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στο τι προσάγγιση έχουμε στην Ιταλία για το ε, leader. Ποια είναι τα δυνατά σημεία, ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά και τελικά έχω και κάποιες προτάσεις για το ε, τι εφαρμογή θα μπορούσαμε να κάνουμε σε σχέση με την ΚΑΠ μετά το 2020. Σε αυτήν την διαφάνεια μπορείτε να δείτε ε, το σύνολο των ε, ομάδων τοπικής δράσης και βλέπουμε τι αφορά την του, του, του, τους σπόρους από τα διάφορα ταμεία και κυρίως από το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου. Και από εδώ μπορείτε να δείτε το ότι οι πρώτες 10 χώρες ε, παίρνουν 75% από το σύνολο αυτών των ομάδων. Και άρα 18% οι υπόλοιπες 18 χώρες έχουν το υπόλοιπο 25% των ομάδων διορθώνει ο Οπότε από εδώ φαίνεται στην συνέχεια πώς έχουν διατεθεί οι πόροι ε, σε σχέση με το leader. Είναι δηλαδή το 6,9% του συνόλου των πόρων όσον αφορά τις δαπάνες του προπολογισμού. Επίσης, να δούμε τώρα στη συνέχεια το πώς ε, έχουμε προσεγγίσει το leader, τι γίνεται στην πράξη, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια είναι τα μειονεκτήματα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την περίοδο προγραμματισμού στο μέλλον. Έχουμε πάνω από 200 τέτοιες ομάδες που έχουν αναγνωριστεί και τους έχουν διατεθεί ένα δις 200 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ δηλαδή 5,8% των πόρων από το Ταμείο Ανάπτυξη τη Πέθρου και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι θέντες ε, πόροι, έχουν αυξηθεί και οι ομάδες. Και όπως θα δούμε, έτσι, έχουμε κάποιες ε, δυσκολίες. Θα μπορούσαμε να τις ε, ξεπεράσουμε με διορθωτικές κινήσεις. Η δε πολιτική της ε, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης γίνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περιφέρεια. Και βλέπουμε εδώ ότι είμαστε στο 5,8% όσον αφορά τους ε, πόρους που διατίθενται. Βλέπουμε σε ποιες περιφέρειες έχουμε ε, περισσότερες σπόρους, σε ποιες λιγότερο ανάλογα με το χρώμα και επομένως συνολικά βλέπουμε πώς γίνεται η απορρόφηση των πόρων στην Ιταλία, των πόρων του Ταμείου του Ταμείου Ανάπτυξης Τώρα, ε, στην Ιταλία έχουμε πάνω από 60% των ομάδων που καλύπτονται από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και βλέπουμε ότι υπάρχει όμως μία συνέχιση στο, στη χορήγηση των πόρων και έχουμε επαναχρηματοδότηση όσον αφορά την διαχείριση. Οι διαπάνες είναι αρκετά υψηλές, ούτως ώστε να λειτουργούν οι ομάδες τοπικής δράσης. Και από το και από τις ομάδες που αναγνωρίζονται 13% είναι σε καινούργιο ε, μέρη που δεν είχαν προηγουμένως καλυφθεί από το Λίντερ. 6,1 εκατομμύρια ευρώ τώρα βλέπετε ότι έχουμε πάει ε, και βλέπετε πώς έχει γίνει η διαφοροποιημένη πρόοδος. Γενικά μπορεί να δείτε ότι εδώ σε αυτή την διαφάνεια τι καθυστέρηση, τι υστέρηση έχει υπάρξει όσον αφορά τις δαφάνες που αφορούν την προσέγγιση του Λίντερ που είναι στο μη 19. Δηλαδή, όσον αφορά το σύνολο των πόρων, μιλούμε για 1,2 δις ευρώ. Και ε, από αυτά τώρα έχουμε φτάσει στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις του παρελθόντος. Οπότε έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και μία εικόνα για το σύνολο της Ευρώπης. Και ο μέσος όρος έχει φτάσει στο 18,35% όσον αφορά για το μέτρο 19. Αυτές είναι οι δαπάνες. Βέβαια ε, υπάρχει και μία απορρόφηση κάποιων από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξη της Υπέθρου. Επίσης μπορούμε να δούμε εδώ ε, τι ισχύει για όλη την Ιταλία για να δούμε πόσο έχει προχωρήσει κάθε ε, περιοχή της Ιταλίας και βλέπουμε ότι κάποιες ε, περιφέρειες έχουν μεγάλη στέρηση όσον αφορά την ε, απορρόφηση. Βλέπετε τώρα και την ε, αριθμητική ανάλυση για το ίδιο φαινόμενο, τι γίνεται για το μέτρο 19, τι γίνεται για το σύνολο ανά περιφέρεια. Ε, επίσης βλέπουμε πόσες ομάδες τοπικής δράσης είναι σε κάθε ε, περιφέρεια της χώρας και στη συνέχεια βλέπουμε μία σύγκριση για αυτό το σημαντικό μέτρο όσον αφορά τους νεοεσερχομένους νέους γεωργούς. Και βλέπουμε ότι στις περισσότερες περιφέρειες έχουμε λιγότερο ποσοστό ε, από τις ε, ε, διατεθέντων πόρων από όσο όσον αφορά τις ομάδες τοπικής δράσης. Και αυτό αποτελεί μια δυσκολία ούτως ώστε να καλυφθούν όλες οι αιτήσει αυτών των προσώπων. Τώρα ε, είπαμε ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε φτάσει στις 30.000 αιτήσει. Και Υπάρχουν προβλήματα επομένω για την υλοποίηση όλων των μέτρων. Και μπορεί να δείτε τώρα τι γίνεται όσον αφορά την ε, δημοσιονομική εκτέλεση, τι γίνεται για την παλια περιοδο περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, που υπήρχε δυσκολία στην εύρυνση του συστήματος όσον αφορά τους όρους που έχουν διατεθεί. Και το 20% των δαπανών είναι κόστος λειτουργίας. Ε, πρόκειται για πόρους που αφορούν τη γεωργία και οι παρεμβάσεις των ομάδων τοπικής δράσης δεν αφορούν ε, την ε, γεωργία και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έχουμε κάποια διαδικασία επιλογής ομάδων τοπικής δράσης που είναι περίπλοκες. Πρόκειται για υπέρμετη γραφειοκρατία. Τα είπαν και οι προλαλήσαντες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει απλούστευση στην διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά τα συμπεράσματα για να μην υπερβώ το χρονικό όριο, από πλευρά Κοπακοζέκα είπαμε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν το περιθώριο να αποφασίσουν το πώς θα διαθέσουν τα κονδύλια στα πλαίσια του Λίντερ. Και να μπορεί ο καθένας να αποφασίσει επί τη βάση των ιδιομορφιών του. Να μην υπάρχει υποχρέωση να δεσμεύσουν, να διαθέσουν αυτό το 5% τα κράτη. Μπορούν να συμμετέχουν όμως και άλλα ταμεία στην υπόθεση αυτή, όπως το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά τους κοινού στόχους. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει απλούστευση και ελπίζουμε ότι έτσι θα γίνει και τέλος θα πρέπει να δούμε το πώς θα γίνει η μείωση του κόστους λειτουργίας, γιατί θα γίνει με τα μέτρα τα οποία αφορούν τη γεωργία. Σας ευχαριστώ. Ρικάρντο, εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Μίλησες ακριβώς 10 λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα για να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον η συνεδρίαση, ως Πρόεδρος θα ανακατέψω την σειρά των ομιλητών που θα ακολουθήσουν. Και ο κύριο Σότο θα μιλήσει πριν τον κύριο Λούκε. Αν συμφωνείτε. Συμφωνείτε. Ωραία. Οι συνάδελφοι συμφωνούν. Thank you uh, uh, very much for inviting me to this very Σα ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση. Εγώ θα σας παρουσιάσω τη δική μου προσωπική σκοπιά. Θα αντλήσω κάποια συμπεράσματα από την προσωπική μου πείρα. Ε, καλύπτοντας όλη την περίοδο του Λίντερ, Ήμουν από τους πρώτους ε, διαχειριστές του Λίντερ στην Ισπανία και τώρα είμαι το σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και συμμετέχω σε πολλά δικτύα καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Λίντερ. Θα αντλήσω κάποια διδάγματα από το παρελθόν και θα προτείνω και κάποιες ε, συστάσεις για το μέλλον. Βλέπετε μία σύνοψη του περιεχομένου. Έχω πολλές διαφάνειες ε, στο PowerPoint. Ε, μερικές θα τις αφήσω κατά μέρους για να περιοριστώ στο δεκάλεπτο. Καταρχήν, ποια είναι τα βασικά στοιχεία τη συζήτηση. Καταμέτρηση των αποτελεσμάτων είναι το ένα και δεύτερον, διευκόλυνση των αποτελεσμάτων. Πώ θα καταφέρουμε να έχουμε αποτελέσματα πέραν του ε, να τα καταμετρήσουμε και δεν είναι αντιφατικέ αυτέ οι δύο ανάγκε. Θα καλύψω, όπω σας είπα, όλη την περίοδο του Λίντερ. Όπω βλέπετε από αυτό το διάγραμμα, έχουμε δύο σημαντικές ε, αυξήσεις του Leader. Καταρχήν από, τη, από τα σπάργανα του πέρασε σε φάση πιλωτική, μετά από το δεύτερο Leader περάσαμε στο ενισχυμένο Leader, Leader Plus και περάσαμε από την εφηβεία του Leader στην ε, πρώιμη ενήλικη ζωή του. Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα άλματα στην ανάπτυξη του ε, Leader. Από το να περάσει στην παιδική ηλικία στην εφηβεία δεν ήταν μεγάλο το άλμα, αλλά το μεγάλο ποιοτικό άλμα έγινε ε, με το mainstreaming του Λίδερ, τη συνεκτίμησή του σε διάφορες πολιτικές, τότε ήταν που ε, αναπτύχθηκε σημαντικά. Ε, ήμουν ο διαχειριστής του σχεδίου του Cherry Valley, της κοιλάδας των κερασιών. Δεν θυμάμαι καν πώς ήταν το, η κατάσταση τότε. Δεν είχαμε τοπικά προϊόντα, δεν είχαμε τοπικό τουρισμό. Αυτά ήταν ανήκουστα τότε. Είμαστε πραγματικά στον πάτο της ανάπτυξη και βλέπετε μερικά στοιχεία. Καταρχήν τουριστικά καταλήμματα από 150 περάσαμε στα 2.000. Τοπικά προϊόντα δεκαπλασιάστηκαν, Εξαγωγέ κερασιών εξαπλασιάστηκαν, 150 νέες επιχειρήσεις, πάνω από 1.000 νέες θέσει εργασία δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν. Και το σημαντικό σημείο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν οφείλονται όλα αυτά στο leader, αλλά το leader σίγουρα έδρασε ε, καταλητικά για, για να διευκολύνει αυτή τη μετάβαση. Χρειάστηκε να βρούμε τους επιχειρηματίες, να τους εκπαιδεύσουμε, να φέρουμε τον κόσμο σε επαφή, να τους στηρίξουμε. Κάτι τέτοιο δεν θα είχαν συμβεί με τέτοιο τρόπο και με τέτοια ταχύτητα χωρίς το Λίντερ. Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας του. Καταρχήν, οι επενδύσεις που κάναμε στα κοινωμένα σχέδια και στη δημιουργία ικανοτήτων Επίσης, συνδυάσαμε δέσμες μέτρων ε, ήπιας και σκληρής φύσης, ηλισμικού και λογισμικού. Ελαστικότητα. Ήταν η ε, διαγωνισμή πολύ ελαστική και τα κριτήρια προσαρμόστηκαν στις τοπικές ανάγκες. Ε, ταχύτητα, άμεσες πληρωμές, προκαταβολές και επίσης πολυταμιακή προσέγγιση από το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Κοινωνικό Ταμείο και το Αναπτυξιακό Ταμείο. Οπότε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε. Αυτό είναι το πρώτο μου μήνυμα. Ό,τι λειτουργεί να το κρατήσουμε. Και βλέπετε εδώ μια γραφική παρουσίαση πώς, του πώς λειτουργούν τα πράγματα. Καταρχήν είχαμε κάποια κινούμενα σχέδια για τις ε, ομάδες τοπικής δράσης και χρησιμοποίησαμε διάφορα ελαστικά εργαλεία προκειμένου να καταλήξουμε σε ιδέες και να τις διαβρύνουμε σε επόμενη μεταγενέστερη φάση. Και περάμε στο παρατηρητήριο του Λίδερ. Συμμετείχα και σε αυτό. Δύο βασικά στοιχεία από αυτή τη διαφάνεια. Καταρχήν αναγνωρίσαμε κάτι που ισχύει ακόμη, ότι το Λίδερ ήταν και είναι ακόμη το μόνο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου τα θεσμικά όργανα λένε στον τοπικό πληθυσμό σας εμπιστευόμαστε και να σχεδιάσετε τις στρατηγικές και να επιλέξετε τα προγράμματα. Πολύ σημαντικό αυτό το βήμα πάνω από 3.000 ομάδε συμμετείχαν και αυτό είναι τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Δεύτερον, φάνηκε ξεκάθαρα ότι το Leader δεν ήταν ένα απλό μηχανισμό ε, για την ε, δημιουργία πρότυπων μέτρων. Ήταν ένα ολόκληρο εργαστήριο και έτσι θα πρέπει να το, εξετα... να το θεωρήσουμε ω εργαστήριο που στήριξε τη μετάβαση ε, για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Επίσης, ένα εργαστήριο και για την τοπική δημοκρατία. Και κάτι πολύ σημαντικό στις παρούσες συνθήκες, εργαστήριο για τη διασύνδεση ε, των ε, τοπικών πληθυσμών με το, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εγώ θα σας ε, παρουσιάσω τις εμπειρίες μου από την Αλία, γιατί επεκτείναμε το Λίντερ και στις παράκτιες ζώνες. Και η σημασία της εμπειρίας αυτής ήταν τεράστια, γιατί δημιουργήθηκε μια στενή σχέση με τους αλληλείς, με τους ψαράδες. Άρχισε το Λίντερ να διευρύνεται σε θέματα Αγροτική ανάπτυξη, καλύπτοντα και την αλία και με το Φάρνετ, επικεντρωθήκαμε σε συγκεκριμένο τομέα και να εντάξουμε το τομέα σε συγκεκριμένη επικράτηση, συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, η διασύνδεση τομέα και περιοχής. Τώρα, στην επόμενη φάση, όπως σας είπα, το 2007 είχαμε ένα σημαντικό ποιοτικό άλμα. Διπλασιάστηκε το Λίντερ, επεκτάθηκε στις αγροτικές περιοχές και είχαμε μια πολύ σημαντική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου τότε που είπε ότι το Λίντερ δεν εφαρμόστηκε με τρόπο που να αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία του. Δεν εφαρμόστηκε με τέτοιο τρόπο. Και μάλιστα από όρια αυτή τη σημαντική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ήταν μια ε, μεγαλύτερη προσπάθεια όλων των ε, Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να προτείνουν τον κανονισμό κοινών διατάξεων και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές με λεπτομεριακές συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στενήθηκε πολλά συμπεράσματα και πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου. Δυστυχώς όμως ε, δεν ήταν τα αποτελέσματα τα αναμενόμενα, γιατί διαπιστώθηκαν πολλοί αγαθές προθέσεις σε όλα τα επίπεδα, αλλά δυστυχώς προτάθηκαν και επιπλέον περιπλοκές. Και μάλιστα σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση στο κόκκινο βλέπετε ότι ε, 4 πέμπτα 700 περίπου ομάδες τοπικής δράσης ερωτήθηκαν και 4 πέμπτα δήλωσαν ότι η γραφειοκρατία περιόριζε την ικανότητά τους να εφαρμόσουν το leader. Πραγματικά σοκαριστικό αυτό το στοιχείο. Και εδώ με τις ε, ε, εφαρμογές και, την, και τις αρχές του leader, διαπιστώνουμε ότι, ότι από τις σημαντικότερες αρχές για την ανταπόκριση στο, στις νέες προκλήσεις, η πολυτομεακή προσέγγιση, η στήριξη της καινοτομίας και της συνεργασίας, αυτές οι αρχές είναι οι πιο δυσεφάρμοστες κατά τη γνώμη των ομάδων τοπικής δράσης. Και βλέπετε τα στοιχεία που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πίνακα και βλέπετε τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Είναι τεράστιες οι διαφορές. Και βλέπετε ότι σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση καινοτόμων λύσεων, οι ομάδε τοπική δράση θεωρούν ότι στα, καλύτερα στα χειρότερα κράτη-μέλη στα χειροτερα είναι 11%, ε, στα καλύτερα 100%. Τεράστια διαφορά στην εφαρμογή από 11 μέχρι 100%. Οπότε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση του leader στο μέλλον. Καταρχήν θα πρέπει να επιτρέψουμε στο, με, στο leader να κάνει αυτό που κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κάθε παράδειγμα είναι και μία ιστορία. Ε, και έχω links στις διαφάνειές μου που σας παραπέμπω σε αυτές τις ιστορίες. Στο Βέλγιο δημιουργήσαμε τοπικά οικοσυστήματα τροφίμων στη Γερμανία, βιοενεργειακά χωριά, στην Ουαλία, πράσινη κυκλική οικονομία, στη Γαλλία, ο ψηφιακός κόσμος είναι μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Επίσης, ε, στηρίξαμε πρωτοβουλίες για την ευρυζωνικότητα στα πλαίσια των έξυπνων χωριών. Αυτές και επίσης κάποιες εφαρμογές για την καλύτερη κινητικότητα. Ήδη οι ομάδες του Leader διευκολύνουν ε, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και δίνουν το αναρτήριο λάκτισμα για την προώθησή τους. Εμείς θα πρέπει να επιτρέψουμε στο leader πραγματικά να κάνει το, τη δουλειά, να υλοποιήσει την αποστολή του. Και βλέπετε από το τελευταίο σεμινάριο στην Αυστρία που είχαμε, ποια είναι τα χρήσιμα για τις εγχειριστικές αρχές. Να δοκιμαστούν ε, νέες προτάσεις, ε, να χρηματοδοτηθούν σχέδια λογισμικής φύσεως, ε, να, χρηματο... να βρεθούν κονδύλια για επενδύσεις ηλισμικής, ηλισμικού ε, χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, ε, συμφωνώ με κάποια σχόλια ότι θα πρέπει να αποτυπώσουμε καλύτερα την προστιθέμενη αξία και να καταμετρήσουμε. Αριστερά έχουμε τους συμβατικούς δείκτες ε, που ε, καταμετρούν τα επιτέγματα του Λίντερ και βλέπετε και μια δημοσκόπηση που κάναμε επί τόπου. Ε, επισκεφτήκαμε εννέα αυστηριακά σχέδιο και από τα εννέα σχέδια μόνο εννέα θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν. Γιατί δεν είναι τα σχέδια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά κοιτάξτε τα άλλα επιτεύγματα των σχεδίων αυτών. Ε, ώρες ε, εθελοντισμού. 344 εταίροι, νέες ομάδες 250, διασυνδέσεις με άλλα σχέδια 48. Βλέπετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Leader. Αυτά θα μπορούσαμε να τα αποτυπώσουμε καλύτερα για να φανεί θέμενη αξία. Και εκεί ίσως θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και να έρθω σε κάποια συμπεράσματα και συστάσεις που έγιναν από τους ε, συμμετέχοντες στο τελευταίο σεμινάριο που κάναμε στο δίκτυο Ευρωπαϊκής, ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης στο ρούς της Αυστρίας. Καταρχήν, ε, χρειαζόμαστε καλούς κανόνες, κατάλληλους όμως για την υλοποίηση των στόχων μας. Οπότε το πρώτο είναι να ε, διακρίνουμε τους κανόνες του leader από τους υπόλοιπους κανόνες και οι βασικοί κανόνες ε, εφαρμόζονται άσχετα με τις ιδιαιτερότητες. Επίσης, ε, να έχουμε κάποια συστήματα που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του leader και οι κανόνες να είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργούν ε, ικανότητες, θα προετοιμάζουν το έδαφος για μικρά σχέδια, συλλογικά σχέδια, πιλωτικά, πειράματα. Γιατί στη θεωρία όλα επιτρέπονται, αλλά στην πράξη δύσκολα υλοποιούνται. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να γίνουν όλα αυτά στις διάφορες χώρες να προλιάνουμε το έδαφος και να τα διευκολύνουμε. Τρίτον, να συμπεριλάβουμε τις ομάδες τοπικής δράσης στη χάραξη των κανόνων, στη θέσπιση, στο σχεδιασμό των κανόνων. Θα πρέπει όλο το σύστημα από το χαμηλότερο επίπεδο, το περιφερειακό, το εθνικό, το ευρωπαϊκό, όλα τα επίπεδα να συνεργάζονται στη χάραξη των κανόνων, ώστε οι κανόνες να ανταποκρίνονται στους στόχους που θέλουμε να υλοποιήσουμε, να είναι κατάλληλοι για την υλοποίηση των στόχων. Τέταρτον, αυτό που ακούσαμε και από τους προλαλήσαντε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε ε, στα αποτελέσματα για το leader, να αναπτύξουμε κατάλληλους δείκτες για να αποτυπώσουμε και να παρακολουθήσουμε την προστιθέμενη αξία, την ουσιαστική προστιθέμενη αξία του leader και τέλος δεν αρκούν οι κατευθυντήρες γραμμές και καθοδηγήσεις και τα έγγραφα η ερμηνεία. Δεν αρκούν καν οι κανονισμοί. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια παρακολούθηση της εφαρμογής επιτόπου. Το είπε ο κύριος Πράιορ για τη σημασία των αγροτικών δικτύων. Θα πρέπει να υπάρχουν ανταλλαγές απόψεων, ε, ε εκπαίδευση, κατάρτιση για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε κύριε Σότο με συγκίνησε το πρώτο παράδειγμα που δώσατε ε, για τα κεράσια και μάλιστα δύο μέλη της Επιτροπής μας ε, σίγουρα είναι υπέρ αυτής της ε, επιλογής το ότι μας βολεύει το cherry picking το cherry picking δεν το καταλαβαίνω το έχει παρεξηγήσει η κυρία Μέ γι' αυτό μην το πείτε το σχόλιο μου ο κύριος Ρόμπερτ Λούκης τώρα έχει το λόγο Ε, είμαι ο Ρόμπερτ Λούκε, προέρχομαι από την Αυστρία και θα μιλήσω στα γερμανικά. Είμαι σύμβουλος ε, και έχω προβεί σε πολλές αξιολογήσεις ε, προγράμματα αγροτική ανάπτυξης του Λίντερ αλλά και άλλων ειδών προγραμμάτων σε διάφορα πλαίσια και σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να συζητήσω ένα πολύ σημαντικό ζήτημα μαζί σα. Το Leader δημιουργήθηκε ω μια κοινοτική ε, πρωτοβουλία ε, τη δεκαετία του 1990. Υπήρχαν αυτές οι επωνομαζόμενες κοινοτικές ε, πρωτοβουλίες τότε που είχαν φτάσει ως τις 13 και εστίαζαν σε τρία τίνα αυτές οι πρωτοβουλίες. Ε, καταρχήν στην εξέβρεση εξατομικευμένων, εξειδικευμένων λύσεων σε ό,τι αφορούσε συγκεκριμένα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης ε, σκόπευαν στο ε, ε, να πειραματικά να διερευνηθούν νέοι τρόποι διακυβέρνησης και επίσης είχαν ως σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας, know-how, την πρόθεση της συνεργασίας και ούτω καθεξής. Ε, leader κατάφερε να επιβιώσει. Το 2007 είχε γίνει βέβαια αυτή η μεγάλη προσπάθεια του mainstreaming, της ένταξη δηλαδή όλων αυτών των στοιχείων στα, ε, στις ευαστικές πολιτικές, αλλά το leader κατάφερε να διατηρήσει και τον ακέραιο χαρακτήρα του, γιατί το ε, leader αποτελεί ταυτόχρονα και θεωρία ανάπτυξη, αλλά και μέθοδο ανάπτυξη και μέτρο ανάπτυξης. Και γιατί το Λίντερ κατάφερε ε, να επιβιώσει ακριβώς ως ένα υποδειγματικό πρόγραμμα. Καταρχήν επειδή αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο για την προώθηση των κοινωνικών προ... Ε, καινοτομιών. Ε, γιατί ε, δεν δίνει προτεραιότητα σε τεχνολογικού χαρακτήρα καινοτομίε, γιατί αυτές οι καινοτομίε ε, είναι τυφλές εντό εισαγωγικών απέναντι στη βιωσιμότητα. Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργείται και έρχεται στην αγορά, είτε αυτό είναι για παράδειγμα στον τομέα των μέσων κοινωνική δικτύωση, είτε στον τομέα τη τεχνητική νοημοσύνη, αλλά δεν σημαίνει αυτή η καινοτομία ότι θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα για όλου. Αν όμω δούμε τώρα τον ορισμό ε, τη κοινωνική καινοτομία, θα διαπιστώσουμε ότι στο τέλο αυτή η κοινωνική καινοτομία εμπλουτίζει, βελτιώνει, ενισχύει την κοινωνική ζωή όλων γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάτι ως κοινωνική καινοτομία. Άρα λοιπόν το leader αποτελεί ακριβώς ένα τέτοιο πλαίσιο προώθησης ειδικότερα κοινωνικών καινοτομιών από τις οποίες κοινωνικές καινοτομίε ναι μπορούν να προκύψουν και τεχνολογικού χαρακτήρα, τεχνολογικο-οικονομικού χαρακτήρα καινοτομίε. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ε, ότι το leader εστιάζει στην ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής και κατά συνέπεια λαμβάνει υπόψη την διαφορετικότητα, την πολυμορφία των επιμέρους φορέων. Άρα λοιπόν εδώ ο βασικός φορέας είναι ομάδα της τοπικής δράσης. Και περνάω εδώ στις βασικές αρχές του Λίντερ καθώς ε, το Λίντερ αποτελεί μια μέθοδο και ακριβώς μία μέθοδο η οποία συνδυάζει τα διαφορετικέ αρχές του leader, δηλαδή η ε, λήψη υπόψη των ιδιωτεροτήτων το ονόμα, το, η ε, τοπική εταιρική σχέση, η πολυτομιακή προσέγγιση, η ολοκλήρωση σε κοινωνικό επίπεδο, η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ε, τοπικών περιοχών και η δικτύωση, η δημιουργία δικτύων. Και υπάρχει και μια όγδοη αρχή, η οποία ε, ε, αποτελούσε μέρος των 7 τότε αρχών ε, το 1990, δηλαδή η συμμετοχή στη διαχείριση και την χρηματοδότηση. Αυτό, αυτή λοιπόν η αρχή είχε εξαφανιστεί στη συνέχεια, αλλά επανεμφανίστηκε στο CLLD. Γιατί στο CLLD προβλέπεται ακριβώς ότι η ομάδα τοπικής δράση είναι η αρμόδια σε ό,τι αφορά και το σχεδιασμό, αλλά και την υλοποίηση τη στρατηγική αγροτικής ε, ανάπτυξης και θεωρώ πως πραγματικά αυτή η αρχή, η επιχειρησιακή δηλαδή αρχή, είναι η 8η αρχή. Γιατί αν υπάρξει παράβαση αυτής της 8ης επιχειρησιακής αρχής, τίθενται ε, ένα αμφιβόλο και οι υπόλοιπε 7 επιχειρησιακές αρχές. Ε, ποια είναι η θεωρία ε, του leader, σε ποια θεωρία βασίζεται αυτή η θεωρία είναι σημαντική για μα, για του αξιολογητέ των προγραμμάτων του Λίντερ. Δηλαδή, εξετάζουμε πάντα ποια είναι η λογική ενό προγράμματο Leader και γι' αυτό ακριβώ καλούμαστε σε αυτέ τι περιπτώσει να τεκμηριώσουμε, να αποδείξουμε ότι η λογική ενό προγράμματο ακολουθεί ακριβώ την θεωρία του Λίντερ. Και βέβαια με βάση τα όσα διαπιστώνουμε προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να εκλεπτύνουμε, να, να, να εξελίξουμε ακόμα περισσότερο μια θεωρία. στους κύκλους λοιπόν των αξιολογητών των προγραμμάτων του Λέντερ έχει καταστεί σαφές ότι το, η, βασική αρχή που καθιστά το ε, leader επιτυχημένο είναι ακριβώς ε, και η ε, μέθοδος ε, που ακολουθεί και για την αξιολόγηση του. Γιατί βέβαια διαφοροποιείται και από αυτό που συμβαίνει για παράδειγμα σε άλλα είδη αξιολογήσεων. Γιατί αυτό το input με το output είναι το ίδιο το input και το output είναι τα ίδια. Δηλαδή, όταν επενδύω στην συνεργασία, λαμβάνω συνεργασία. Όταν επενδύω στην συμμετοχή, τότε το output, το αποτέλεσμα είναι και πάλι συμμετοχή. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα γίνεται μετρήσιμο μόνο στο επίπεδο των γενικότερων αποτελεσμάτων, τη απόρριας δηλαδή αλλά αυτό αποτελεί πρόβλημα μόνο σε περίπτωση όπου κανείς προβαίνει σε αξιολογήσεις ε, με πολύ περιορισμένο τρόπο, όπου δηλαδή προβαίνει απλά σε μετρήσεις μηχανιστικού χαρακτήρα. Η αξιολόγηση αποτελεί μια επιστήμη, μια εφαρμοσμένη επιστήμη, η οποία βασίζεται σε αρχές μικροοικονομικές αλλά και μακροοικονομικές ή οικονομετρικές ε, θεωρίες και αντίστοιχες εφαρμογές. Ε, στο Leader όμως, αν δούμε Ε, καταρχήν ε, σε τι βασίζεται η λογική της παρέμβασης θα διαπιστώσουμε ότι Έχουμε καταρχήν την τοπική στρατηγική ανάπτυξη ε, και την εφαρμογή της ε, μέσω ε, project Επίση επίσης έχουμε την ευαισθητοποίηση και δημιουργία ικανοτήτων μέσω των ομάδων τοπικής δράσης από την πλευρά των φορέων και η διαμόρφωση και η διαχείριση των εργαλείων ακριβώς χρηματοδοτικής υποστήριξης. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία μπορεί κανείς να διαπιστώσει κατά πόσο το leader είναι επιτυχημένο ή όχι. Και το εξετάζουμε σε σχέση με τρει τομεί. Καταρχήν, σε ποιο βαθμό ένα πρόγραμμα leader εμπλουτίζει το κοινωνικό κεφάλαιο και αυτό μπορεί κανεί να το μετρήσει, ω κοινωνικό δηλαδή κεφάλαιο. Και αποτελούν, δηλαδή εδώ ε, συντίθεται από στοιχεία τόσο ηθικού ε, ε, χαρακτήρα, για παράδειγμα όπως η αλληλεμιβαία εμπιστοσύνη, αλλά και διαστάσεις της δικτύωσης. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι η ικανότητα διακυβέρνησης, ε, δηλαδή η ποιότητα συνεργασίας ε, των δημοσίων, ε, των ιδιωτικών αρχών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε ό,τι αφορά την εκτέλεση δημοσίων ή μάλλον κοινωνικών καθηκόντων. Και ο τρίτος τομέας των αποτελεσμάτων είναι τα καλύτερα ε, project, ε, δηλαδή τα πιο συμμετοχικά, τα πιο ισορροπημένα, τα πιο βιώσιμα project. Αλλά σε ό,τι αφορά την αντικειμενική μέτρηση αυτών των κατηγοριών, μόνο η τρίτη μπορεί να μετρηθεί με καλύτερο τρόπο. Εγώ έχω ε, συμμετάσχει σε τέτοιου είδου μελέτε κόστου αποτελέσματο και έχω διαπιστώσει όταν κανεί προβαίνει στην αξιολόγηση ενό προγράμματο leader και διαβάζει μία σειρά από αριθμούς εδώ, προβαίνει σε μία σύγκριση για παράδειγμα με project εκτός leader και διαπιστώνει ότι τα προγράμματα leader τελικά οδηγούν στην μόχλευση, αν θέλετε, στην κινητοποίηση περισσότερων ιδιωτικών ε, ε, επενδύσεων, πέραν και των όσων μπορούν να ε, δημιουργήσουν σε επίπεδο εθελοντικών πρωτοβουλίων. Επίσης, δημιουργούν περισσότερη δυνατότητα αποδοχής των σχετικών υπηρεσιών, καινοτόμων υπηρεσιών και επίσης διαπιστώνουμε ότι τα ίδια κονδύλια στο πλαίσιο ενός ε, προγράμματος ε, ε, Leader επιτυχάνουν περισσότερα, υψηλότερο ποσοστό. Για παράδειγμα, στο δικό μου κρατήριο του Ζάξεν, Ε, περιλαμβάνει, ε, ε, χρησιμοποιεί το 41% των κοντιλίων για το Leader και αναφέρει ότι αναφέρεται από εκείνη την πλευρά ότι εκείνο που πραγματικά τους έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι βλέπουν πραγματικά να υπάρχουν πολλά αποτελέσματα γιατί ακριβώς είναι και πολύ προσεκτικοί και παρακολουθούν επακριβώς τον αντίκτυπο των κοντιλίων που αξιοποιούν. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ανησυχεί τους αξιολογητές το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να μετρήσουν. Δηλαδή οι ανθρωπιστικές επιστήμες προσφέρουν τις απαραίτητες ε, ε, ε μεθόδους. Ε, για παράδειγμα, outcome harving, realist evaluation, outcome mapping ε, ε, και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες μεθοδολογίες, απλώς δεν εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής. Ωστόσο, είναι δυνατόν να μετρήσουν λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν βασιζόμαστε στο ότι το leader θα έπρεπε να εφευρεθεί αν δεν υπήρχε ήδη. Και αυτό βέβαια καταδεικνύεται και από το γεγονό ότι ο αριθμό των ομάδων τοπική δράση αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Δηλαδή παρόλο, παρόλα τα προβλήματα που ανέφερε, ε, ε, ε ανέφερε και ο συνάδελφο Χόισλερ, ε, υπάρχει πραγματικά προστιθέμενη αξία και ε, σπάνια προσεγγίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον απλό πολίτη τόσο πολύ όπως μέσω του προγράμματος Leader. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ε, έχουμε πάντοτε κατά νου τις αρχές του Leader ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και την παρακολούθηση του Leader. Ας δώσουμε λοιπόν το κατάλληλο ε, επίσημο πλαίσιο ε, και για την αξιολόγηση του leader, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ταυτόχρονα ε, και την, τα αντίστοιχα εργαλεία στις αρμόδιες αρχές εφαρμογής. Και θα πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω την δικτύωση και σε εθνικό και διά περιφερειακό επίπεδο, γιατί εκεί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα πραγματικά και τέλος θα πρέπει να επεκτείνουμε και να διευρύνουμε τη μέθοδο ε, του Λίντερ στο πλαίσιο του CLLD σε ό,τι αφορά και άλλες ιδιαίτερες περιοχές όπως για παράδειγμα τις αστικές, περιαστικές, παράκτιες και ούτω καθεξής. Κάτι τέτοιο μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε περισσότερα διδάγματα ε, και σε περισσότερη εμπειρία από την οποία μπορούν να υποφεληθούν όλοι οι υπόλοιποι σε σχέση με τα όσα έχει επιφέρει το Leader στις αγροτικές ε, περιοχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, θα αφήσω τώρα τις μεγαλύτερες ομάδες, τον κύριο Τσέλερ και Χόισλινγκ και θα δώσω το, το λόγο στον κύριο Φλάναγκαν, στην πιο αριστερή ομάδα. Μια σύντομη ερώτηση για τη συνεισφορά σε σχέση με αυτά που είπε ο Ιταλός εκπρόσωπος. Είπατε 20% της διοίκησης. Αρχικό ποσοστό ή γενικό. Ή μόνο για την Ιταλία ισχύει αυτό το 20%. Άλλες ερωτήσεις. Οπότε ερωτώ τους πανελίστες μας. Θέλετε να απαντήσετε, ίσως με τη σειρά που εκφωνήσετε και τις ομιλίες σας. Αν και η ερώτηση ήταν μάλλον για τον Ιταλό εκπρόσωπο. Κύριε φλάνα, θα είχατε την καλοσύνη να επαναλάβετε την ερώτηση, αν δέχεστε τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Ναι, αναφερθήκατε στο 20% για τη διοίκηση. Αυτό ισχύει μόνο για την Ιταλία ή είναι γενικό στοιχείο, γενικό ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Yeah, please. Um, I think it's I think it's really important to um... είναι, είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ διοίκησης και απορρόφησης. Running costs. το, τα animation, το κόστος λειτουργίας animating the, the, the, the territory. Um, so I, can't, com- I don't have figures on... Άλλο γινόμενα σχέδια, άλλο διοικητικές δαπάνες. Όχι, δεν έχουμε εδώ κάποιο συγκριτικό πίνακα. Μήπως έχει κάποιος άλλος. Uh, in, in recent evaluation and studies, I always... Ανέκαθεν. Θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι πήγε το κατόφλι στο 25%. Έτσι ορίζει ο κανονισμός. αν κανείς μιλήσει με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται το Leader, λένε ότι όλα αυτά απορροφούνται, εξαφανίζονται λόγω της ακραία γραφειοκρατίας και του χαρτοβασιλείου. Δεν είναι εύκολο να τα αποφύγουν. Οπότε θα ήθελα να υπάρχει περιθώριο πέραν από την ανάπτυξη των σχεδίων και της πλαισιωστής τους. Να έχουν το χρόνο για να υπάρχει ευαισθητοποίηση, ενημέρωση για αυτά ακριβώς. Δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν το περιθώριο, γιατί έχουν πάρα πολλά να κάνουν λόγω γραφειοκρατίας. Α, πολύ ζωντανή συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος και ο κύριος Τσέλερ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Τσέλερ. Άκουσα προσεκτικά όλα όσα είχαν να πούν οι δικοί μας. Εγώ εργάζομαι στην Περιφερειακή Επιτροπή και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, όχι στην Επιτροπή Γεωργίας. Και το πάγιο ερώτημα για το Λίντερ είναι στα προγράμματα του. Ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος. Και ακούσαμε από τους ειδικού ότι πολλοί εμπλεκόμενοι θεωρούν ότι υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Οπότε και τα προγράμματα κολλάνε. Όλοι μας θα πρέπει να σκεφτούμε επομένως πώς θα πλουστευτεί η κατάσταση. Αλλιώς θα χάσουμε αξιοπιστία και δεν θα μπορέσουμε να την ανακτήσουμε. όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό άλλο να με την διαχείριση της υπαίθρου. Αλλά άλλο το πρόγραμμα των ανάπτυξης της υπαίθρου και άλλο οι άμεσες πληρωμές. Ο γενικός κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει αυτούς τους ε, γεωργούς που έχουν τις ενισχύσεις. Να ευθυγραμμίζονται τα προγράμματα και θα πρέπει να είναι συμβατά τα προγράμματα της γεωργίας με τα προγράμματα της ανάπτυξης. Τι λέτε. Ευχαριστούμε κύριε Τσέρα, λέει ο Πρόεδρος. Βλέπω ότι δύο από τους καλεσμένους μας ζήτησαν το λόγο. Κυρία Μποτέλιο πρώτη. Ε, για το 20% των διοικητικών δαπανών που ερωτήθηκε. Αυτό το θέμα του 20% των διοικητικών δαπανών αφορούν ε, λειτουργία, ε, ε δαπάνες λειτουργίας ε, αλλά και ενθάρρυνσης των περιοχών. Επίσης, ε, τα τοπικά επιτελεία δημιουργούν και θέσει απασχόληση, ειδικευμένε που απασχολούνται στι αγροτικέ περιοχέ και αυτό είναι μια ευκαιρία για να παραμείνει κανεί στην Ήπεθρο. Γιατί εκεί που εντοπίζονται τα προβλήματα θα πρέπει να βρίσκουμε τι λύσει σε τοπικό επίπεδο. Μπορούμε να συμφωνούμε να διαφωνούμε για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, αλλά το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης χρήζει μεγαλύτερη υποστήριξη για να έχουμε μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη. Και αν βγει από τα ΕΔΕΤ, δεν θα αναλαμβάνονται υπόψη τρει πυλώνε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα υπάρχει μεγαλύτερο κατακαιρματισμό. Γι' αυτό είμαστε υπέρ τη πολυταμιακή προσέγγιση με διαχείριση σε τοπικό επίπεδο από ένα συντονιστικό φορέα στο οποίο συμμετέχουν οι ομάδες τοπικής δράση Ο κύριο Φατζόνε για να απαντήσω στην ερώτηση για το 20% για την Ιταλία τον έφερα και ως επιτοπλίστων αυτά οι πόροι διατίθενται για την γεωργία. Και βέβαια Υπάρχουν οι δαπάνες ε, λειτουργίας, οι δαπάνες ε, της λειτουργίας. Οπότε ως κόπα κοντζέκα θα θέλαμε να υπάρξει ε, περισσότερη διάθεση από αυτούς τους πόρους, περισσότερα χρήματα για τη Γεωργία. Και τώρα θα κάνω κάτι ασυνήθιστο. Θα ξαναγυρίσω στο πρώτο πάνελ και θα δώσω το λόγο στην κυρία Λόριτς Χόφμαν, αλλά για ένα λεπτό μόνο. Και θα είστε και τελευταία ομιλήτρια επ' Έχετε τεράστια ευθύνη λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την τεράστια ευθύνη που μου αναθέσατε. Καταρχήν, γιατί η πολιτική αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να εξακολουθεί να καλύπτεται από το κανονισμό περί κοινών διατάξεων και για τα υπόλοιπα ΕΔΕΤ, όπως ισχύει τώρα. Θα είμαι σαφής. Η ε, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ε, συνδέεται με την ε, κοινή γεωργική πολιτική για να εξασφαλίσουμε δρομολόγηση των κονδυλίων στις αγροτικές περιοχές. Θέλουμε περισσότερα χρήματα να δαπανώνται για τις, να δαπανώνται για τις αγροτικές περιοχές. Δυστυχώς όμως οι πόροι είναι επενιχροί και προέρχονται κυρίως από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα έχει ένα γενικότερο πλαίσιο στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα πια της ΚΑΠ. Θέλουμε μια γενική στρατηγική για να βλέπουμε τι συμβαίνει γενικώ στη Γεωργία ε, και άλλες δραστηριότητες ή υποδομές στις αγροτικές περιοχές και προτείναμε μια ειδική προσέγγιση που θα στηρίζεται στις επιδόσεις και γι' αυτό χρειαζόμαστε στενή σχέση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα για να αναπτύξουμε αυτή την ιδέα. Και πάνω από ένα χρόνο ε, εξετάσαμε τη δυνατότητα της συμπερίληψης του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και συμφωνήσαμε με τους συναδέλφους σε άλλες γενικές διευθύνσεις τελικά ότι δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο γιατί θα έπρεπε να επιτρέψουμε πολλές παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις και η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης ε, μόνο για μερικά τμήματα του CPR θα ήταν κατάλληλη. Οπότε θέλ, προτιμήσαμε να την αποκλείσουμε πλήρως από το δημοσιονομική διαχείριση και το ελέγχου σε περίπτωση που θα είχε μπει στο κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να αξιοποιούμε ό,τι μας ε, εξυπηρετεί από το κανονισμό περί κοινών διατάξεων στο leader. Και εκεί παίρνουμε αυτά που μας εξυπηρετούν από το CPR και πολλές άλλες έννοιες και τα εφαρμόζουμε αμέσως στον κανονισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και συνεχίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα ταμεία και μας ενδιαφέρει αυτή η πολυταμία και προσέγγιση και τα κράτη-μέλη στα σχέδιά τους για την ΚΑΠ θα πρέπει να μας πούν με τι μηχανισμούς εξασφαλίζεται συνοχή με την υπόλοιπα ταμεία. Γιατί το έδαφος είναι κοινό, είναι κοινό το πεδίο όλων των ταμείων και αυτό θέλουμε να γίνεται σωστό έργο. Ακόμη και αν η πολιτική αγροτική ανάπτυξη δεν καλύπτεται πλήρω από τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, αλλά από μερικέ μόνο διατάξει του. Ευχαριστώ. Έχω και άλλα δύο καθήκοντα. Το ένα είναι διαδικαστικό, να εγκρίνουμε δηλαδή τις συστάσεις των συντονιστών μας. Ήδη σας μοιράσαμε τα συμπεράσματα της πρωινής συνεδρίας των συντονιστών και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε έγγραφη μορφή. Και αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις θα θεωρηθούμε ως συγκεκριμένα τα πρακτικά τις συστάσεις μάλλον των συντονιστών της Επιτροπής Άκρη. Ο κύριος Φλάναγκαν. Θα ήθελα να σημειωθεί στα πρακτικά ότι σχεδόν δεν έχει απομείνει κανένας για να εγκρίνει τη στάση των συντονιστών. Α, συγγνώμη, υπάρχει και μία άλλη συνάδελφος. Η απαρτία σας λέει κάτι. Η έννοια της απαρτίας σας λέει κάτι. Γιατί στην τοπική μας κοινότητα χρειαζόμαστε απαρτία για να λάβουμε κάποιες αποφάσεις. Αλλιώς ακυρώνεται η συνεδρίαση. Θα ήθελα κύριε Φλάναγκα να σας ενημερώσω ότι είστε κοντά στο να χρησιμοποιήσετε το πυρηνικό όπλο. Αποθαρρύνουμε όλους τους ευρωβουλευτές να κάνουν έλεγχο απαρτίας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε δημόσια κρόση. Τώρα από ότι η απαρτία που έχουμε είναι αρκετή. Η προσέλευση μάλλον που έχουμε είναι αρκετή. Εκτός μικροφώνου. You There are too many micros here. <laughs> so basically, dear experts, colleagues, and the court. Ακούσαμε λοιπόν τους εμπειρογνωμονές μας από το ελεκτικό συνέδριο, από τους ε, τοπικούς ε, φορείς οι δύο μα λοιπόν ε, κοινοβουλευτικέ επιτροπέ αποφάσισαν να διοργανώσουν από κοινού αυτή την ακρόαση, γιατί εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συχνά θέλουμε να έχουμε μια καλή σφαιρική επισκόπηση σε ό,τι αφορά ειδικότερα τι ε, πολιτικέ μα αγροτικέ ανάπτυξη. Ε, και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τις κριτικές της τοποθετήσεις σε ό,τι αφορά τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ένωση και φυσικά σε αυτό το πλαίσιο εξετάζει και το κόστος της διαχείρισης η η Επιτροπή Γεωργίας συχνά παρουσιάζεται ως ε, η Επιτροπή που έχει ε, τις υψηλότερες δαπάνες υπό την αρμοδιότητά της ε, και η οποία ασχολείται περισσότερο με τους γεωργούς και με τις σχετικές πολιτικές. Και βέβαια ο στόχος είναι πάντοτε να λαμβάνουμε διδάγματα από το παρελθόν και να βελτιώνουμε το μέλλον. Όπως βλέπουμε σε αυτόν τον τομέα των αγροτικών περιοχών δηλαδή υπάρχουν ακόμα πολύ σοβαρά προβλήματα όπως υποαπασχόληση, όπως ελλειπείς υπηρεσίες και ούτω Άρα λοιπόν υπόψη και την κύραση του πληθυσμού πληθυσμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει τρόπου ε, προκειμένου να παραμείνει ο πληθυσμό στι αγροτικέ περιοχέ, χωρί όμω υπερβολική διοικητική επιβάρυνση. Εγώ προέρχομαι από μια τέτοια περιοχή ε, και μπορώ να φανταστώ ότι ε, είμαι ο νεότερο που κατοικεί στο χωριό μου, παρότι είμαι κι εγώ μιας προχωρημένη ηλικία. Άρα λοιπόν η σημερινή ακρόαση μας βοηθάει να αντιληφθούμε λίγο ε, καλύτερα ε, το πώς ε, μπορούμε να δώσουμε συνέχεια στις αυτές τις πολιτικές. Τα δύο πάνελ παρουσίασαν διαφορετικές διαστάσεις και ίσως το βασικότερο δίδαγμα που έχουμε αντλήσουμε είναι ότι το leader έχει πραγματικά τη δυνατότητα να δημιουργήσει συνέργειες σε τοπικό επίπεδο δημιουργώντας πολύτιμα project τα οποία σε διαφορετική περίπτωση δεν θα δημιουργούνταν. Όπως είπε ο κύριος Λούκης, εάν δεν υπήρχε το leader θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η συνεδρίαση ολοκληρώνεται εδώ. Ευχαριστώ τους πάντες και ιδιαίτερα τους διαμενείς.